Good afternoon. Sui tempi dobbiamo essere molto perché poi è buono. Ecco, ecco, ecco. Good afternoon everybody. Good afternoon. Welcome. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρία ή μάλλον μεσημεριανή συνεδρία. της ημερίδας που από το πρωί έχει ξεκινήσει και που εντάσσεται στο πλαίσιο του πακέτου για τη μετανάστευση. Και τώρα το δεύτερο μέρος αφορά τις ενδοϊπηρεσιακές μεταθέσεις. ICT όπως τους λέμε, τους μετατιθέμενους ενδοϊπηρεσιακούς. Σαγητής είναι ο κύριος Γιακολίμ. Θα του δώσω το λόγο να μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασία του. Μετά θα ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου καθώς και την εισηγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης που σας υπενθυμίζω τη βάση του άρθρου 50 του αστερικού μας κανονισμού συνεξετάζει την ε, πρόταση αυτή της Κομισιόν. Λοιπόν, ποιοι συνοδεύουν τον κύριο Γιακολίνο στο βήμα. Καταρχάς κάποιος πολύ γνωστός σε όλους μας, ο κύριος Στέφανο Μανσερβίση, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Καλώς ήλθατε για μια ακόμη φορά κύριε Μανσερβίση. Επίσης η κυρία Βίβιν Βιντάση, Βάνταση, που ήταν και το πρωί μαζί μας, στην πρωινή συνεδρία. Είναι σύμβουλος της Μονάδας Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ξέρουμε ότι η Ουγγρική Προεδρία αυτή τη στιγμή ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνάδελφός μας Λίσα για Κονσάρη, συγγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης. Καλώς ορίσατε και εσείς. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σας υπενθυμίσω. Ήδη από τώρα σας το λέω έχουμε πρόβλημα με το χρόνο και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πολλοί από εμάς ναι έχουμε να, να προλάβουμε τις πτήσεις μας. Φεύγουμε για τις διακοπές του Πάσχα, που όπως ξέρετε πλησιάζει. Και επειδή θα χρειαστεί να βιαστούμε για το αεροδρόμιο, καλό θα ήταν να μην καθυστερήσουμε και γι' αυτό πρέπει συνέχεια να έχουμε το ρολό στο μυαλό μας. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Γιακολίνο. Καλησπέρα σα. Ε, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω όλου σα ε, τους συναδέλφους και καλωσορίζω βέβαια και όλους όσοι θα ακολουθήσουν μετά από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Πρόκειται για πρόταση οδηγίας την οποία σήμερα θα σχολιάσουμε. Θα ασχοληθούμε με τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει Αυτά τα οποία θα ακούσουμε σήμερα το απόγευμα συσχετίζονται με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Κυρίως εργαζόμενους που προέρχονται από τρίτες χώρες και οι οποίοι ήδη έχουν ενταχθεί μέσα σε ιδιωτικές δομές εργασίας, μέσα σε ε, επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για το πώς οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε δομέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια την επιχείρηση και αυτά βάσει μια οδηγία, η οποία την προηγούμενη χρονιά παρουσίασε η Επιτροπή ως μέρος ενός πακέτου που αφορά στη νόμιμη μετανάστευση. διαφάνεια και ενιαίες ρυθμίσεις στην αγορά. Αυτά είναι απαραίτητα προαπαιτούμενα για την οδηγία, η οποία οδηγία έχει ως στόχο να ρυθμίσει τις μεταναστευτικές ροές, αυτές οι οποίες εμφανίζονται στην αγορά εργασίας, ε, έχοντας ε, κατά κύριο λόγο ως στόχο τους ε, τα προσόντα τα οποία προέρχονται από τον πολιτισμό του καθενός. Αυτή η οδηγία αφορά τις ε, διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που είναι σαφείς, χωρίζονται με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο. Θα αναφερθώ σε αυτά αργότερα. Εδώ γίνεται λόγος για τους ε, μάνατζερ, για τους ε, πτυχιούχους, γίνεται λόγος για επαγγελματίες, εξειδικευμένους επαγγελματίες, ε, κυρίως ε, επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν ε, σημαντικά και με σοβαρό τρόπο στην οικονομική βιωσιμότητα της ενιαίας αγοράς. Πρόκειται για την ευκαιρία που μπορεί να προσφέρεται στους εργαζομένους αυτούς και στις οικογένειές τους έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα της ε, οικογενειακής επανασύνδεσης. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο εξετάστηκε από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Είναι ένα έγγραφο ε, το οποίο βεβαίως και πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Σήμερα το πρωί Είπαμε ότι θα πρέπει ενδεχομένω να γίνει μια αναθεώρηση τη συμφωνία ε, του Σέγγεν λόγω των μεγάλης, της, της μεγάλης πίεσης των ε, μεταναστευτικών ρεών που δεν έχει σταματήσει. Εχθές θα ξέρετε ότι είχαμε 700 μετανάστες οι οποίοι προέρχονται όχι μόνο από την Βόρεια Αφρική αλλά και από την υποσαχάρη Αφρική ε, έφτασαν αυτοί στην ε, Λαμπεντούζα και αποβιβάστηκαν με τη βοήθεια της ε, ακτοφυλακής της Ιταλίας. Το θέμα λοιπόν των μεταναστευτικών ροών είναι καθοριστική σημασίας και για τον πολιτιστικό διάλογο και για τον διαθρησκευτικό αλλά και διότι αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του ε, ισχύοντος οικονομικού συστήματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι η οδηγία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν μπορούμε σε πολιτικό επίπεδο να αρνηθούμε τη σημασία που έχουν οι μηχανισμοί ελέγχου έτσι ώστε να αποφύγουμε τον εκφυλισμό, να αποφύγουμε το ενδεχόμενο της ε, κατάχρησης. Ε, οφείλουμε να έχουμε ένα εργαλείο που θα μας ε, επιτρέπει να μην υπάρχει εκφυλισμός της νόμιμης μετανάστευσης. Θα μετατραπεί η, μετα... η νόμιμη μετανάστευση σε κάτι τελείως διαφορετικό. Βεβαίως και τα κράτη-μέλη και εκείνα πρέπει να συνδράμουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιδείξουν αλληλεγγύη. Αυτά είναι θέματα που έχουν συζητηθεί επανειλημμένα. Την τελευταία φορά συζητήθηκαν στις 4 Απριλίου κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Στρασβούργου. Εμείς ε, επιθυμούμε να υπάρχει ε, μια ταχεία αλλά ενδελεχής ε, έρευνα της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμούμε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προτάσεις που θα κατοτεθούν και εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος όπως ε, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μεταβατική περίοδος δεν θα βοηθήσει στο να ρυθμίσουμε ή να εξηγιάνουμε καταστάσεις οι οποίες ήδη υφίστανται. Θεωρούμε ότι το εργαλείο αυτό, δηλαδή η μεταβατική περίοδος ε, ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τις ε, οικονομικές επιπτώσεις, κάτι που αναφέρεται σε μια έρευνα που έκανε η Επιτροπή, αυτό θα μπορούσε να διοχετεύσει τους ε, εργαζόμενους σε, στην αγορά εργασίας, τους ε, επαγγελματίες υψηλού επίπεδου, οι οποίοι για, τρεις ή για τρία ή τέσσερα χρόνια θα μπορούσαν να εργαστούν στον ε, τομέα αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει θα υπάρχουν ενιαίες ρυθμίσεις και διαφάνεια στην αγορά εργασίας και στα κράτη-μέλη. Ε, στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να λαμβάνεται επίσης υπόψη ότι η ευελιξία είναι και αυτή ένα θέμα που και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ε, το θέμα των ε, ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων είναι ένα θέμα που, για το οποίο ε, πολλοί επιθυμούν να συμβάλλουν, όπω είπε και ο πρόεδρο, και εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφέροντα απλά και μόνο το εξή. Θεωρούμε ότι αυτό το θέμα μπορεί να ενταχθεί μέσα στην στρατηγική του 2020 που αφορά στην βιώσιμη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η δική ε, παραμονή. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στον ανταγωνισμό και αυτό εκμεταλλευόμενοι ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα αντιμετωπιστεί ως κοινοτικό δυναμικό. Και εδώ προβάλλεται λοιπόν το στοιχείο της ε, κοινοτικής αντιμετώπισης. Ολοκληρώνω την ε, ομιλία μου ευχόμενος ε, στους ε, υπόλοιπους εισηγητές να συνεργαστούμε για το άρθρο 50 και στο πλαίσιο του άρθρου 50 ίσως τελικά κατορθώσουμε να επιτύχουμε μια πραγματικά σοβαρή και αξιόπιστη συνεργασία και ελπίζω και σε ένα αρκετά εύλογο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε και σας ευχαριστούμε επίσης και που σεβαστήκατε το χρόνο που σας είχαμε διαθέσει για να μας βοηθήσετε να ε, διεξάγουμε αποτελεσματικά τη συζήτηση. Ο πρώτος είναι ο κ. Μαλτσερβίση, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Doesn't? Eh, okay, okay, it's fine. Well, thank you, thank you, Mr. Um, President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ιακολίνο για την παρουσίαση και για την ε, δουλειά που κάνετε. Θα πρέπει να πω ότι συζητώντας αυτή την πρόταση σήμερα μπορεί να φαίνεται κάπως παράξενο γιατί εδώ μιλάμε για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ανησυχούμε για τα όσα συμβαίνουν ιδιαίτερα στην Νότιο Μεσόγειο όμως είναι σημαντικό επίσης να τα τοποθετήσουμε όλα αυτά σε ένα πλαίσιο που ε, από το 2005 η Κομισιόν έχει υποδείξει ποια θα έπρεπε να είναι η ακολουθητέα πολιτική ώστε να ρυθμιστεί η μετανάστευση που είναι προς το συμφέρον μας. Και γι' αυτό αυτή η οδηγία, όπω αυτή που συζητείτε σήμερα για του εποχιακού εργαζόμενου είναι ένα από τα τελευταία τμήματα αυτής της, ε, ε, αυτού του οράματος που θεσπίστηκε το 2005. Γιατί διαρκώ μιλάμε για τους μακροπρόθεσμους ε, κινδύνους, βράχοι πρόθεσμου συγγνώμη, κτλ. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ήπειρος ε, διαρθρωτικής μετανάστευση και ότι στη στρατηγική μας για ανάπτυξη είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε σωστά την μετανάστευση ώστε να τα καταφέρνουμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της, του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτό, όπως λέω συχνά, είναι κατανοητό όσον αφορά την δημογραφική συρρήκνωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Είναι ένα γενικό πλαίσιο αυτό. Λιγότερο κατανοητό, ωστόσο, είναι, ή λιγότερο σαφές είναι, ε, είναι ο λόγος για την ποιότητα της εξέλιξης αυτής, τις ανάγκες πρέπει να καλύψουμε για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε θέση τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε προς το καλύτερο το δυναμικό της εσωτερικής μας αγοράς. Αυτή η οδηγία ακριβώς σε αυτό το ε, τμήμα αναφέρεται, το τμήμα που, εξερτά, ε, που εξετάζει την μετανάστευση ως κάτι που είναι προς το συμφέρον μας. Προς το συμφέρον μας όχι μόνο γενικόλογα, αλλά αντιμετωπίζει τις δυνατότητες καλύτερης εκμετάλλευσης εσωτερικής αγοράς, διότι αυτή η οδηγία αποτελεί έναν τρόπο για να ε, μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς μας είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θεωρείται εμπόδιο, αλλά αντιθέτως είναι απαραίτητο συστατικό μιας οικονομίας που είναι ανοιχτή ανοιχτή στις επενδύσεις και μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτό για να δημιουργήσει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα με βιώσιμο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πρέπει να δει κανεί αυτή την πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή να το δει κανεί ω μια αντίθετη τάση από την ε, έννοια κλειδί της σημερινής συζήτησης, αλλά ελπίζω πως θα συνειδητοποιήσουμε όλοι πως πρόκειται για το δικό μας συμφέρον. Γιατί είναι για το δικό μας συμφέρον, γιατί σε όλα τα έγγραφα που έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ακόμα και αν δεν έχουν εγκριθεί, αποτελούν τμήμα του προβληματισμού για το πώς θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσε να είναι πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Οικονομία, ε, αναγνωρίζεται ότι πρέπει να επενδύσουμε στις γνώσεις, στην προηγμένη τεχνολογία και στην καινοτόμα οικονομία, για να τα πούμε έτσι πιο σύντομα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να είμαστε ελκυστικοί όσον αφορά τους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που αποτελούν τμήμα μέλη μιας εταιρεία που ήδη είναι εγκατεστημένη εδώ ή που υπολογίζει να εγκατασταθεί εδώ πράγμα το οποίο αποτελεί τμήμα της ελκυστικότητας ενιαίας αγοράς μας για ε, τις επενδύσεις. Μιλάμε δηλαδή όχι για κάτι που δημιουργεί νέα μετανάστευση, αλλά για κάτι το οποίο ρυθμίζει την κίνηση ατόμων που αποτελούν τμήμα ενός συνόλου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αυτή δεν είναι μια οδηγία που έχει στόχο να αυξήσει τη μετανάστευση, ακόμα και αν αυτή είναι νόμιμη, αλλά θέλει να επιτρέψει στις εταιρείε να κινούν μέσα στους ομίλους τους ε, ανθρώπους που είναι ε, υψηλά ιστάμενοι υπάλληλοι, managers κτλ. Ε, και είναι μέλη του, είναι μάλλον υπάλληλοι ενό ομίλου και πρέπει να μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα. Αυτό είναι ο στόχος και το όριο αυτής της οδηγίας. Και γιατί δεν ήταν απαραίτητο να νομοθετήσουμε από αυτού, γιατί... Αυτή είναι φυσικά η πρώτη ερώτηση. Γιατί να νομοθετήσει κανείς σε σχέση με τις ενδο υπηρεσιακέ μεταθέσει. Καταρχήν, οι πολυεθνικέ εταιρείε, οι εταιρείε που επενδύουν εδώ, χρειάζεται να φέρουν προσωπικό από αλλού. ώστε να μπορούν να του τοποθετήσουν καταλήλω στα διάφορα τμήματα της εταιρεία. Τώρα, αν αυτή πρέπει να είναι μια ενέργεια που θα δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα μεγαλύτερη με ομαλό τρόπο, θα πρέπει, θα ήταν σκόπιμο να διευκολύνουμε αυτές τις μετακινήσεις ή όχι. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμή υπάρχει ένα παζλ από νομοθεσίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν επιτρέπει ακριβώς αυτή την ομαλή μετακίνηση των υψηλά ειστάμενων και δικευμένων ανθρώπων που είναι υπάλληλοι πολυεθνικών εταιριών που οργανώνουν παραρτήματα, θηγατρικές κτλ. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα μιας ενιαίας αγοράς ελκυστικής και γι' αυτό είναι και είναι απαραίτητο μέσω μιας νομοθεσίας να βρούμε ένα, να φτιάξουμε μάλλον ένα ε, ισότιμο πεδίο. Μιλάμε για υψηλά εστάμενο προσωπικό, είπαμε μάνατζερ, ε, διευθυντές κτλ. οι οποίοι μετατίθενται μέσα στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής εταιρείας, ενός ομίλου. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους γνώσεις που δεν υπάρχουν και δεν είναι διαθέσιμοι ε, στην ίδια εταιρεία επιτόπου. Και άρα στόχο δεν έχουμε να δημιουργηθεί ένας μόνιμος τρόπος για αυτούς τους ανθρώπους να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος μιας άλλου μέσου της μπλε κάρτας. Απλώς ε, θέλουμε ο κόσμος αυτός που είναι ούτως ή άλλως ανήκει σε μια εταιρεία να μπορεί να παραμείνει επί προσωρινής βάσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι λοιπόν ότι η διαμονή προβλέπεται για περιορισμένο χρόνο, για περιορισμένη διαμονή, προσωρινή διαμονή αυτός είναι δευτερεύον στόχος. Η πρώτο στόχος είναι ελκυστική, ελκυστικό πεδίο για επενδύσεις, περισσότερη δηλαδή οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να τα καταφέρουμε όλα αυτά, ποια είναι τα βασικά εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. τα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέλη ενός μιας εταιρείας. Πόσο καιρό θα μου πάρει ας πούμε να πάρω άδεια παραμονής. Πρέπει να οργανώσουμε ένα, μια γρήγορη, ένα γρήγορο τρόπο. Μια εταιρεία που πρέπει να φέρει λοιπόν τον κόσμο της πρέπει όχι μόνο να ανταποκριθεί σε διαφορετικές νομοθεσίες αλλά και σε απρόβλεπτες ε, ε περιστάσεις. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια διαδικασία σύντομη και μια ενιαία άδεια που καλύπτει την παραμονή και την άδεια εργασία. Δεύτερον, λένε αυτοί οι άνθρωποι να εντάξει να το κάνω. Εγώ να έρθω εδώ και να δουλέψω και σαν μέλος κάποιου, κάποιο ιδρύματος, ας πούμε, να πάω στην ΕΑ στη Μάλτα που μόλις δημιουργήθηκε, αλλά θέλω να φέρω και την οικογένειά μου. Και άμα δεν φέρω την, μπορώ να φέρω την οικογένειά μου, δεν θα έρθω. Άρα λοιπόν δεύτερος στόχος είναι να επιτρέψουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και γρηγορότερο τρόπο την επανένωση την οικογενειακή. Τρίτο στοιχείο, μας βλέπουν ως μια νέα αγορά. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει είσοδο για μια χώρα, εκεί που βρίσκεται το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να ρυθμίσουμε πώς μπορεί κανείς, αυτοί οι άνθρωποι μάλλον, να μετακινούνται στην ενιαία αγορά για να μπορούν να δουλέψουν έτσι όπως οργανώνεται η δουλειά της εν λόγω εταιρεία. Και τελευταίο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη με βέλεκτο τρόπο ποιοι είναι οι αριθμοί που χρειάζονται και καθορίζονται από τα κράτη-μέλη. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με το βασικό στόχο τη οδηγία. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν αριθμητικά στοιχεία. Είναι μια αρχή τη συνθήκη αυτή. Αν λοιπόν Θα πρέπει να μπορεί η εταιρεία να ξέρει τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, σε ενιαία αγορά. Καλύτερη και γρηγορότερη λοιπόν πρόσβαση στην ε, παγκόσμια σκηνή για να γνωρίζει κανεί τι πρέπει να κάνει. Και αυτό ισχύει όχι μόνο. Ε, αυτό είναι προ όφελο όχι των εταιρεών, αλλά και προ όφελο τη Ευρώπη. Όχι από αποτέλεσμα μόνο της δραστηριότητας αυτής της εταιρείας αλλά και της παρουσίας των ανθρώπων αυτών που ε, δημιουργούν γνώση, δημιουργούν ειδικευσή σε συγκεκριμένους τομείς και είναι αυτό ωφέλιμο για όλους μας. είναι ένα είδος ε, αγοράς που δεν καλύπτει όλο τον κόσμο εννοείται Μιλάμε για περίπου 60.000 ανθρώπους που είναι παρόντες σε ένα σύστημα το οποίο είναι κατακαιρματισμένο για την ώρα και που εμπίπτουν ε, αυτές 60.000 αυτές κατηγορίες. Και έχουμε επίσης αριθμούς που διαφέρουν σε διάφορα κράτη-μέλη. 4.500 στη Γερμανία, 3.000 στις κατοχώρες, 2.000 στη Γαλλία, 1.000 στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Σύμφωνα με τις ε, στατιστικές του ΩΣΑ, αυτού του είδους οι μεταθέσεις αφορούν ε, το 4% των παγκόσμιων μετακινήσεων και της μετανάστευσης. Μεγάλος ο αριθμός δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος μετακινείται μέσα σε αυτού του είδους τους ομίλους και τις εταιρείε. Μιλάμε για ειδικευμένους ανθρώπους που φέρνουν μαζί τους γνώσεις, είναι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι, είναι καθορισμένοι και έτσι αποφεύγονται και οι καταχρήσεις. Έχουμε χώρες όπως το, το Ηνωμένο Βασίλειο όπου ε, αυτές οι μεταθέσεις αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο τη μετανάστευση, τη μεταναστευτική κίνηση. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε από την άποψη τη πραγματική προστιθέμενη αξία, εθνικότητα για παράδειγμα. Ε, μιλάμε βασικά για Ινδούς, Αμερικανούς, Κορεάτες, Ιάπωνες Κινέζους, όλο και περισσότερους Κινέζους, γιατί όσο οργανώνονται οι κινέζικες εταιρείες ως πολυεθνικές, εγκαθίστανται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία μου παρατήρηση. Αυτοί είναι οι κανόνες που προβλέπουμε, Αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο ε, έχουμε προβλέψει την νομοθεσία. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα φυσικά, αλλά η συζήτηση και ο τρόπος βιοθέτησης ε, μέσω της συναπόφασης φυσικά θα βελτιώσει τα πράγματα. Γι' αυτό και είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Η διαδικασία είναι χρήσιμη για να βελτιωθεί το πράγμα, γιατί θα μπορεί να είχαμε κάνει λάθη. Ε, άνοιγμα λοιπόν. Αλλά ας μην ξεχνάμε το εξής είναι τόσο σημαντικό όσο και η ύπαρξη της ίδιας ενιαίας αγοράς. Η ενιαία αγορά είναι σημαντική όχι επειδή δημιουργεί ισότιμο πεδίο για τις εταιρείε, αλλά και γιατί αποφεύγει αυτή τη τάση που είναι καταστροφική για την οικονομία και για τους ανθρώπους εδώ στην Ευρώπη να δημιουργούν εθνικούς πρωτοθλητές και να πιστεύουν ότι μια χώρα μπορεί να επενδύσει περισσότερο στη γνώση και να είναι καλύτερη και άρα να συμβάλλει περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτό είναι καταστροφικό. αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να απεφευθεί αυτός ο ζημιογόνο ανταγωνισμός. Τη μία φορά τη φορολογία, την άλλη αφορά την ελκυστικότητα, την άλλη το κόστος της εργασίας. Είναι ένας τρόπος ώστε όλοι να υποχρεωθούν να δουν την ενιαία αγορά ως μια πραγματική δοκιμή. Ε, αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε γιατί αυτό θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστεί ο ζημιογόνος ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, στο να δημιουργούν δηλαδή εθνικές καλύτερες συνθήκες με την αυταπάτη ότι θα συμβάλλουν περισσότερο στη δική τους ανάπτυξη. Αυτή είναι η βασική λοιπόν προσέγγιση, βασικές πτυχές και επαναλαμβάνω ότι είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε όλες τις απαραίτητες τροπολογίες για να το βελτιώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Mrs. Σας ευχαριστώ κύριε Μασερβής. Κύριε Βαντάση τώρα, εκ μέρους της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης και για το θέμα των ενδοϊπηρεσιακών μεταθέσεων και το σχετικό σχέδιο οδηγίας. Η Προεδρία μας προσδίδει μεγάλη σημασία στο να ακούσουμε τις απόψεις των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων. Και βέβαια με τα χαράς και εγώ θα σας εκθέσω την κατάσταση πώς έχουν μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η οδηγία των ενδοϊπηρεσιακών μεταθέσεων, όπως ε, είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι ένας άλλος ακρογωνιαίος λήθος για αυτό το πακέτο ε, μέτρων σε σχέση με την νόμιμη μετανάστευση. Θεωρούμε ότι στόχο έχει να προτείνει ένα απλό λειτουργικό σύστημα που θα καταστήσει ελκυστική την Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για το έγγραφο εργασία του και να πω εκ των προτέρων ότι ε, σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων και για τα χρήσιμα συμπέρασματα τα οποία πιστεύω ότι θα αποκομίσουμε στο τέλος της συνεδρίασης αυτής. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω ουγγρικά τώρα. Κυρίες και κύριοι, η Ουγγρική Προεδρία αντιλαμβάνεται πολύ καλά τη σημασία του θέματος αυτού και ιδίως ε, τον αντίκτυπο που έχει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών. Υπάρχει προστιθέμενη αξία στο σχέδιο αυτό το επεσήμανε άλλωστε και ο Γενικό Διευθυντή προηγουμένω. Δηλαδή ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα εναρμόνιση. θέμενη αξία λοιπόν, κοινοί ορισμοί, κοινά κριτήρια υποδοχής, μια πιθανή τουλάχιστον κατ' επιλογή, και ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδίδουν αξία στο σχέδιο αυτό είναι η κινητικότητα. Η κινητικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ομάδα εργασίας για τη μετανάστευση στο Συμβούλιο και γίνονται εντατικές συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος της μεταφοράς, της πρακτικής εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα είναι απλή Μιλάμε για άτομα που μετατίθενται ενδοϊπηρεσιακά, αλλά θέλουμε οι διαδικασίες να είναι γενικώ απλές. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, όπως σας είπα, έχει συζητήσει σε αυτόν τον καιρό, οι περισσότερες από τις οποίες ασχολούνται με το θέμα της κινητικότητας. Στο σχέδιο υπάρχουν διατάξεις για την κινητικότητα. Έχουμε εγκύψει σε αυτά τα θέματα Έχουμε αρχίσει να τα εξετάζουμε και αυτό το οποίο περιέχει το κείμενο προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και για στρατηγικούς λόγους αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα είδος ε, κοινό μοντέλο για την κινητικότητα. Αυτό το έχει αναλάβει η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και με ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι το συνολικό αυτό μοντέλο το στηρίζει και η Κομισιόν. Αυτό το μοντέλο ε, παρτίζεται από δύο πτυχές, αν θέλετε. Αφενός, κινητικότητα μικρών αποστάσεων, οπότε εκεί θα έχουμε μια ταχεία διαδικασία, fast track, και αφετέρου μια ε, πιο παραδοσιακή διαδικασία για μακρών αποστάσεων κινητικότητα. Μια άλλη πτυχή που μας έχει απασχολήσει είναι τα κριτήρια υποδοχής και εισόδου Αυτά τα κριτήρια πρέπει να είναι απλά για τις αρχές που θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία πρώτα απ' όλα. Πρέπει οι αρχές αυτές να είναι σαφές ότι οι υπήκοοι τρίτων κρατών εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας. Ο κύριος Γιακολίνο νωρίτερα μίλησε για καταχρήσεις. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί, άρα πρέπει να είναι σαφής οι διατάξεις οι σχετικές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη είναι όλο το θέμα της άρνησης, εισόδου, της απόσυρσης ή η αιτιολόγηση της μη ανανέωσης της άδεια. Σίγουρα και εδώ πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφείς οι διατάξεις πάλι για να μην υπάρξουν καταχρήσεις και αν χρειαστεί να είναι δυνατή επιβολή κυρώσεων. Γνωρίζω ότι στο έγγραφό του ο εισηγητής δεν αναφέρεται στην πτυχή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω εγώ αυτή την πτυχή, που οποία είναι σημαντική κυρίες και κύριοι. Επίσης στο σχέδιο γίνεται λόγος για τη δυνατότητα κοινών ορισμών. Κατά τις συζητήσεις της ομάδας εργασίας ανέκυψε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν σαφείς, ακριβείς ορισμούς και ακριβώς προς το σκοπό αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η υπηρεσιακό μετατιθέμενο, η οποία εμπίπτουν στο πεδίο τη της θα χαίρουν μια ε, απλή διαδικασία. Αυτό είναι ο στόχο μα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε κι εσεί ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα. Συνεργαζόμαστε στενά και με την ομάδα εργασία για τι κοινωνικέ υποθέσει. Η δική μα ομάδα εργασία μετανάστευση έχει ζητήσει μάλιστα τη γνωμοδότηση τη ομάδα εργασία για τι κοινωνικέ υποθέσει, γιατί νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τη συνέχιση των ε, συζητήσεων. Και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαβουλεύσει. Επιπροσθέτως έχουμε τα δικαιώματα των ε, μετατιθεμένων, δικαιώματα επίσης περί οικογενειακής επανένωσης για τα άτομα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά και προεξέχοντα στοιχεία. Η Ουγγρική Προεδρία προτίθεται να διοργανώσει συζητήσεις και στο μέλλον για τις διατάξεις αυτές. Θέλουμε αυτό που θα προκύψει τελικά να είναι κάτι που θα δίνει μια συνολική γενική εικόνα της κατάστασης. Αυτό είναι σημαντικό για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχουμε υπόψη τα συμφέροντα και των δύο μερών σε αυτό το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ουγγρική Προεδρία, σημειώνουμε τα ε, ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα και τις απόψεις των κρατών μελών, αλλά όχι μόνο. Και τους κοινωνικούς εταίρους ακούμε, παραδείγματος χάρη, προτάσεις ψηφισμάτων, ε, ε, συνεργαζόμαστε και με την πολωνική Προεδρία, την επερχόμενη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει μια συνέχεια στη δράση μα. Επίση, παρακολουθούμε το σύνοικε εξελίξει εξελίξεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι διαπραγματεύσει που λαμβάνουν χώρα εδώ και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά και στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Βαντάση. Α ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια τη Επιτροπή Απασχόληση, την κυρία Γιακονσάρη. Take the floor. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για που οργάνωσε αυτή την ε, συνάντηση, αυτή την ακρόαση, με συγχωρείτε. Διάβασα το έγγραφο εργασία του συναδέλφου του κ. Γιακολίνου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πού Και διάβασε επίσης και τα σχόλιά του και τις παρατηρήσεις του. Είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και η οδηγία ε, θα προσφέρει υπεραξία στην Ευρώπη γιατί πραγματικά χρειάζεται να ε, βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα αυτής της ε, γυράσκουσας υπήρου. Ένα λοιπόν εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας ε, στους μετανάστες ε, ένα καλό σημείο κίνηση είναι αυτή η συζήτηση. Γιατί θεωρώ ότι τελικά συμφωνούμε όλοι στις βασικές απόψεις ε, που εκφράζει αυτή η οδηγία. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις και κάποια σχόλια προς την Επιτροπή ε, και ίσως και άλλοι επιθυμούν να σχολιάσουν, γιατί πέρα από τις ε, θετικές συνέπειες που θα προκύψουν από την οδηγία υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά. Ε, προφανώς λέμε ότι ε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό λοιπόν θα κάνω και εγώ τις ε, ερωτήσεις μου. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι η σχέση, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην οδηγία και τους αισθητή τους ε, ε, εργαζόμενους αυτούς. Αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ε, μετατεθέντες, αλλά δεν ισχύει οδηγία για την περίπτωσή τους. Πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εάν η οδηγία δεν ισχύει για την περίπτωσή τους, τότε γιατί το αναφέρετε. Τη στιγμή που μιλάμε για άτομα που έχουν εργαστεί ακόμα και για τρία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ήταν πιο απλό και σαφέστερο ε, να ισχύει για αυτούς η ίδια νομοθεσία όπως και στους ε, γηγενείς εργαζόμενους. Εάν δεν πρόκειται να εφαρμοστεί οδηγία, ε, θα υπάρξει πρόβλημα στην εφαρμογή της οδηγίας ε, των ε, εσωτερικών ε, μεταθέσεων. Εγώ δεν νομίζω ότι θα καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή της οδηγίας μιλώντας για μεταθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, η οδηγία τη στιγμή είναι ασαφής. Η πρόταση αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ευνοϊκότερους ε, κανόνες ε, ε, στην κατηγορία αυτή των υπαλλήλων από ότι στους απλά μετατεθέντες. Πάντως ε, οι αποσπαστέντες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα από τους ντόπιου. Στην Σερδική 2020 η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλαμβάνεται της, ε, των τοπικών διαπραγματεύσεων. Εδώ όμως η οδηγία έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση, ε, δίνει περισσότερη σημασία στην χώρα προέλευσης και βλέπω ότι εδώ υπάρχει μια σαφής αντίφαση. Πάντως με το να θέλουμε να επιφέρουμε μεγαλύτερη διευκρίνηση φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε ένα αρνητικό, κακό νομοθέτημα. Συμφωνώ με τον κύριο Γιακολίνο ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τους ορισμούς. Τι είναι τελικά εμπειρογνώμονας ε, με πολλά προσόντα. Είναι λιγάκι ασαφής ο ε, ορισμός και μπορεί ε, να επιδεχτεί πολλές ερμηνείες. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Σε αυτή την οδηγία για τους εργαζόμενους ε, που έρχονται από τέτοιες χώρες και βρίσκουν εργασία μέσα από ένα γραφείο ευρέσεως εργασίες ισχύει για αυτούς η σχετική οδηγία ή η οδηγία οι εργαζόμενοι με τη μορφή υπεργολαβίας ε, ποιος είναι αρμόδιος εάν η αλυσίδα υπεργολαβιών περιλαμβάνει διάφορες εταιρείες και τους εργαζόμενους. Και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ε, το καθεστώς των κυρώσεων κατά άποψή μου είναι αρκετά ασαφές. Δεν ε, προβλέπονται στην πρόταση ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου ε, και θα ήθελα να γνωρίζω, να πω το εξής. Εάν η Κομισιόν επιθυμεί να λύσει το θέμα με τη συνεργασία των κρατών μελών, αυτό είναι λιγάκι αφελές. Γιατί το θέμα δεν μπορεί να λυθεί απλά με τη συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και μεγάλες χώρες όπως είναι η Κίνα, παραδείγματο Ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει, δεν φέρει θετικά αποτελέσματα η συνεργασία. Θα ήθελα να πω στον κύριο Γιακολίνο ότι όσον αφορά τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις οικογένειες, την οικογενειακή ζωή ε, και να επιδείξουμε την απαραίτητη ευελιξία. Παρά λοιπόν τις παρατηρήσεις που έκανα προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία με τον κύριο Γιακολίνο και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αυτές τις ε, νομοθετικές διατάξεις και κυρίως για τα ε, θέματα που θα εξετάσουμε στο πλαίσιο της συναρμοδιότητας την οποία έχουμε ήδη ορίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιακονσάρη που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης συναρμόδια με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και τώρα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. κυρία Ρομερα, Ρομερο Λόπες είναι η πρώτη και τη δίνω βεβαίω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θέλω να τον ρωτήσω το εξής. Αυτή την πρόταση οδηγίας που από ό,τι φαίνεται αποτελεί την απάντηση σε μια αναγκαιότητα πιστεύετε ότι πραγματικά θα ανταποκριθεί στους στόχους να ε, είναι η απάντηση σε μια ανάγκη των πολυεθνικών εταιριών που θέλουν να προσλάβουν ε, στελέχη σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η αιτία, ποιος είναι ο βασικός λόγος, ο ουσιαστικός λόγος ε, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη που μπορεί να έχει μια εταιρεία σε κάποιε άλλε χώρες. Αυτοί έχουν λάβει εκπαίδευση εκεί. Όταν μετακινηθούν τώρα αυτοί, η κατάρτιση, η επιμόρφωση, ε, Ποιο την έχει πληρώσει, η ευρωπαϊκή χώρα προέλευση. Και μπορεί να προκύψει το εξή, να πληρώσουν φτωχές χώρες για την μόρφωση, για την εκπαίδευση ε, στελεχών που για λόγου ανταγωνιστικότητα ε, υπό ανταγωνισμού των πολιεθνικών ε, τα στελέχη αυτά θα μετακινηθούν σε μια πιο πλούσια χώρα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο τελικά. Να περνάνε δηλαδή να μετατίθενται εργαζόμενοι από τις πιο φτωχές τις πιο πλούσιες χώρες. Ε, απλά ερώτηση σας κάνω επειδή δεν το γνωρίζω καλά το θέμα Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η πιο βαθιά αιτία αυτής της πρότασης οδηγίας και να ρωτήσω την εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας. Φυσικά και είναι πολύπλοκο το θέμα και επειδή ακριβώς είναι πολύπλοκο θα πρέπει να δούμε τις καταχρήσεις που μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, αν μπορώ να τις πω έτσι και η ορολογία δεν είναι πολύ σαφής. Στελέχη τρίτων χωρών. Αυτά μπορούν να υποκαταστήσουν ε, τοπικούς εμπειρογνώμονες ή τοπικά στελέχη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η εκπαίδευση γίνεται σε, ε, σε τρίτες χώρες, προέρχονται από τρίτες χώρες. Οι πολυεθνικές τελικά τι έχουν αποφασίσει, να μην μετεγκαθιστούν επιχειρήσεις εξοικονομώντας δηλαδή όλο αυτό το κόστος ε, μεταφοράς. Άρα ε, ναι μεν η έδρα των επιχειρήσεών τους είναι στη δική μας την επικράτεια αλλά με εργαζομένου τρίτων χωρών. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό έτσι. Άρα παρά τις προφυλάξεις και τις ρήτρε ε, που περιλαμβάνει στο άρθρο 14 και στο άρθρο 15 το σχέδιο οδηγίας καθώς και σε ό,τι αφορά το παιδί εφαρμογή της, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Μήπως υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό το 4% των εργαζομένων που προτείνουν ως αριθμητικό στοιχείο, ως νούμερο οι πολυεθνικές. Και αν είναι έτσι κατάσταση, αν δηλαδή είναι λίγο αμφίσιμη και θυπλή, αυτό το θέμα της ταχείας διαδικασίας και της επανένωσης των οικογενειών, ποια διαδικασία θα ισχύσει για αυτά τα θέματα. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα δίνουν αυτές ε, τις άδειε για ταχεία επανένωση των οικογενειών. Άρα, εξασφαλίζοντας καλύτερη μεταχείριση στις πολυεθνικές, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Και φυσικά αυτό είναι καλό για την Ευρώπη, αλλά ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και γιατί να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι πολυεθνικές. Το έχει εξετάσει αυτό η Κομισιόν. Now, Mr. Mulder. Μούλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με πολλά από τα όσα είπε ο κύριος Γιακολίνο στο έγγραφο εργασία. Νομίζω πως η οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να τυποποιήσει την ισχύουσα κατάσταση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για το σκοπό για τον οποίο λέει ότι θα χρησιμοποιηθεί. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει η ίδια περίοδος ε, ε, διαμονής ε, αδειοδότησης για τον υπάλληλο, για το στέλεχος και για την οικογένειά του. Διαφορετικά ε, δεν γίνεται. Παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Πρώτον, ποιος είναι ο ορισμός ενός σταζιέρ. Εγώ εντυπωσιάζομαι όταν έχω τα στοιχεία ανεργίας από την Ιρλανδία, την Ισπανία, που λένε ότι κάποιες φορές 40% των ανθρώπων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να βρουν θέση απασχόλησης. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει κάποια υποχρέωση να αναγκάσουμε αυτές τις εταιρείε ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε μαζί τους να πάρουν πρώτα τοπικό προσωπικό πριν να φέρουν από αλλού. Και τέλος, Ενωπημένη προσέγγιση, ναι, για να είναι ευκολότερο για τις εξένες εταιρείε να εγκατασταθούν εδώ και να λειτουργήσουν, να ευημερίσουν εδώ. Όμως τι γίνεται αντιστρόφως, αν εμείς υιοθετήσουμε αυτό το καθεστώς, σημαίνει ότι θα έχουμε τις ίδιες διευκολύνσεις στη ΣΥΠΑ ή στις ε, χώρες BRICS ή οπουδήποτε αλλού ή πώς δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση που ισχύει διεθνώς. Ευχαριστώ. Κυρία Έρμστ. Όπως και κατά το προηγούμενο σχέδιο οδηγίας και εδώ θέλω να υποβάλω το εξής ερώτημα. Ποιος είναι ο στόχος μας, τι κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Δηλαδή ε, προβλέπουμε να υπάρχει μικρή, μεσαία, ε, μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και άλλων προσοντούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη, να καλύψουμε τα κενά με ντόπιου εργαζόμενους. Ε, ποιο είναι το θέμα, πρέπει να σκεφτούμε σε τι ακριβώς αποσκοπούμε με αυτήν την οδηγία. Και επιτρέψτε μου κάποιες ερωτήσεις Θεωρώ ότι το έγγραφο αυτό είναι ασαφές και δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει ε, όσον αφορά τους όρους, τους ορισμούς. Υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός ε, του όρου όμιλος, όρος όμιλος επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο ή υπάρχει διαφοροποίηση. Τι σημαίνει όμιλος και πώς ορίζεται αυτός. Ε, πρέπει να το κάνουμε αυτό για να ξέρουμε για τι επιχειρήσεις μιλάμε. Μετά, ε, εξειδικευμένος εργαζόμενος, ιδιαίτερα προσοντούχος, Πώς ορίζονται και αυτά. Εξειδικευμένος εργαζόμενος είναι κάποιος ε, που έχει κάνει μια ειδική εκπαίδευση και όταν την έχει ολοκληρώσει τότε εμπίπτει και αυτός στην περίπτωση των αποσπάσεων. Ε, όσον αφορά τους σταζιέρ, έγινε μια ερώτηση, αλλά να ξεκαθαρίσουμε τι είναι σταζιέρ, τι είναι εξειδικευμένο εργαζόμενος, τι είναι ιδιαίτερα προσοντούχος. Με τα ενοικιαζόμενη εργασία, πώς ακριβώς ορίζεται στην οδηγία αυτή όταν μιλάμε για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, πώς ακριβώς το φαντάζεστε εσείς. Και το τελευταίο θέμα που έχω ως πάντα είναι η αποζημίωση. Η εξίσωση ε, με ντόπιου που κάνουν την ίδια δουλειά, ε, πώς ακριβώ το σκέφτεστε αυτό. Ε, αυτό είναι πάντα βέβαια το φλέγον θέμα, οποτεδήποτε ασχολούμεθα ε, με, τα, με τις περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν ε, χώρες όπου δεν προβλέπεται ε, διανόμου ο κατώτατος μισθός και οι χώρες που έρχονται από τρι... οι εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες σε χώρες χωρίς κατώτατο μισθό, πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται αυτοί. Ωραία. Πάμε τώρα πίσω ε, στους μιλητές μας ε, για να ακούσουμε αντιδράσεις ε, πρώτα απ' όλα από τον εισηγητή μας, τον κύριο Γιακολίνο. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις παρεμβάσεις και άκουσα και τις ερωτήσεις και νομίζω ότι εκφράστηκαν κάποιες απόψεις που θα πρέπει να τις λάβουμε επαρκώς υπόψη. Ξεκινάμε με αυτά τα τελευταία που είπατε. Παραδείγματος χάρη, αναφερθήκατε στους ορισμούς είπατε και εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχουμε σαφείς ορισμούς γιατί αλλιώς ορισμός ας πούμε του μάνατζερ αλλά ακόμα και για άλλους υπαλλήλους παραμένει γενικός και άμα είναι γενικός δεν ικανοποιεί ε, την κάλυψη των ελλείψεων, κάτι που έχει ως στόχο κυρίως η οδηγία. Ποιος είναι ο στόχος οδηγίας, το είπαμε. Είπαμε να υπάρχει ένα πλαίσιο αναφοράς, ενιαίο πλαίσιο αναφοράς για τις νόμιμες μεταναστευτικές ροές, να συσχετίζονται αυτές με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σαφές. Όσον αφορά τώρα τους ε, αποσπασθέντες ε, εργαζόμενους υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω και συμφωνώ με αυτούς ε, που έκαναν αυτή την ερώτηση. Ο συνάλφος κύριος Μούλντερ αναφέρθηκε στα θέματα της οικογένειας που και αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως και ορισμός ε, και το ίδιο θέμα τέθη από τη συνάδελφο κυρία Γιακονσάρη την οποία και ευχαριστώ για την υποστήριξή της και που μας έδωσε και κάποιες ε, σχετικές πληροφορίες για τους ε, σταζιέρ υποδοκιμή εργαζόμενους εκεί πράγματι πρέπει να εισάγουμε αυστηρότερα κριτήρια για να αποφύγουμε κάποια στρέβλωση του θέματος όσον αφορά τώρα το ανθρώπινο δυναμικό που έχει εκπαιδευτεί σε φτωχές χώρες και κατόπιν εργαζόμενους εργάζεται σε πλούσιες χώρες. Η οδηγία αυτή μιλάει για μεταθέσεις, αλλά αυτό δεν είναι κατ' ουσίαν μεταφορά. Πρόκειται για απόσπαση, πρόκειται για ένα τρόπο χρησιμοποίησης ιδιαίτερα εκπαιδευμένου προσωπικού, δηλαδή άτομα από τρίτες χώρες που δούλευαν εκεί και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ε, θα εργαστούν στην ε, ίδια επιχείρηση αλλά σε κάποια άλλη μονάδα της ε, επιχείρησης ε, που η μονάδα αυτή βρίσκεται σε κράτος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πράγματι ότι πρέπει να υπάρξει κάποια διευκρίνηση και πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συζήτηση με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτό πράγματι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πολύ ωραία. Ε, ο κύριος Μανσερβίση. Ευχαριστώ. Όταν ε, ξεκίνησε η διαδικασία της συναπόφασης, ε, το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει η Κομισιόν είναι να ακούσει, να κατανοήσει και να διευκολύνει. Να κάνουμε δηλαδή προτάσεις που πιστεύουμε ότι είναι αρκετά κατανοητές για να ανταποκριθούμε σε διάφορα θέματα, αλλά έπειτα πρέπει να διευκολύνουμε την κατανόηση και την συμφωνία στην οποία θα φτάσουμε ενδεχομένω ε, ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η συναπόφαση εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το κατανοήσουμε και γι' αυτό και ακούω προσεκτικά για να μπορέσω να συμβάλλω. Εγώ θα έλεγα να επανέλθουμε στην ουσία αυτής της πρότασης. Η πρόταση αυτή δεν θέλει να δημιουργήσει, μάλλον, θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο μηδενικό όσον αφορά την ποσότητα. Είναι μια πρόταση που στόχο έχει να διευκολύνει την οργάνωση του προσωπικού αντίκτυπο όσον αφορά την ποσότητα. να διευκολύνει την μετακίνηση ανθρώπων που εργάζονται μέσα σε έναν όμιλο. Δεν μπορούμε, μπορούμε να μιλήσουμε για την οδηγία αποσπασμένων εργαζομένων όσον αφορά τους όρους, αλλά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ίδια πράγματα γιατί το θέμα είναι διαφορετικό. Μπορεί να μιλήσουμε για δοκιμές τη αγοράς που δεν αποκλείονται σε κάποια φάση αν κάποιο κράτος μέλος έχει αφιβολίε, ιδιαίτερα για να εφαρμοστεί η προτίμηση η ενωτική αλλά δεν ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί τότε αρνούμεθα το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία οργανώνει τη, δουλειά της, τον τρόπο εργασία της. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε κατηγορίες ανθρώπων που πολλές φορές είναι αόριστε. Το κατανοώ αυτό. Είναι πιο αόριστος όταν μιλάμε ειδικά για σταζιέρ, για ανθρώπου που είναι υποδοκιμοί, εκπαιδευόμενοι. Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στο, όσον αφορά το management. Αλλά για εκπαιδευόμενους, ναι, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μετά υπάρχει το τεστ που γίνεται για να εντοπιστεί ποια είναι η λειτουργική σχέση τι υποτίθεται ότι κάνει αυτός ο άνθρωπος σε συγκεκριμένο οργανισμό ώστε να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά σε συγκεκριμένο μέρος. Γιατί αυτό δεν είναι ένα τεστ αγορά, αλλά είναι ένα τεστ που γίνεται για να δούμε αν και κατά πόσο αυτή η μετάθεση είναι σύμμορφη προς το πεδίο εφαρμογή και του στόχου τη οδηγία. γιατί διαφορετικά μπορεί να αποτελεί κατάχρηση. Είναι μια δοκιμή που μπορεί να γίνει με λειτουργικό τρόπο και πρέπει όντω να έχουμε ορισμού. Αν όμω στη διάρκεια τη διαδικασία διαπιστώσουμε ότι μπορεί να υπάρχει κατάχρηση, φυσικά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μα, αλλά η βασική ιδέα είναι η ευελιξία που να μπορεί να ελέγξει την λειτουργία και όχι μόνο το καθεστώς. Άλλη πτυχή είναι ο έλεγχος του ε, απασχόλησης για το περασμένο δωδεκάμινο. Γιατί αποφασίσαμε να το συμπεριλάβουμε εδώ, διότι υπάρχει άλλη μια ρήτρα που συνδέει αυτή την μετάθεση σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο με ένα συγκεκριμένο σχέδιο της εταιρείας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που γίνεται επί τούτου. θα πρέπει να δούμε και πώς θα μεταγραφεί η οδηγία στα κρατημέλια. Είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στην ευελιξία του να, επιτρέψουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα διοργανώσουμε και όλα, να τα ρυθμίσουμε όλα, γιατί θα πρέπει να ρυθμίσουμε τότε και πώς λειτουργεί κάθε εταιρεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, έρχομαστε κάπου στη μέση. Στη μέση να είναι προ όφελο και τη εταιρεία και προ όφελο δικό μα. Το δικό μα όφελο είναι να επιτρέψουμε σε μια εταιρεία που κάνει επενδύσει, και πιθανότατα επενδύει στην Ευρώπη και πιθανά θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση και περισσότερη οικονομική δραστηριότητα που με τη σειρά του θα δημιουργήσουν και άλλε θέσει απασχόληση, να μπορεί να λειτουργήσει σωστά χρησιμοποιώντα του πόρου τη προ αυτό το σκοπό και χρησιμοποιώντα αυτού του πόρου με αυτέ τι διευκολύνσει για να μπορεί κανεί να μπει στην Ευρώπη, να δουλέψει, να μείνει και να είναι και σε καλύτερη κατάσταση οικογενειακή κτλ δημιουργήσει μια καλύτερη κατάσταση με ανθρώπους που μπορεί να είναι ειδικευμένοι, ναι, μένα, αλλά να ωφεληθούν και από όλα αυτά. Φυσικά θα πρέπει να, να, μην επιτρέψουμε να παρακαυθούν νομοθεσίες ή να στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός. Όμως, η αναφορά στην οδηγία περί αποσπάσεων ακριβώς γι' αυτό γίνεται, για να αποφευχθεί η ενδεχόμενο, ενδεχόμενος του ανταγωνισμός με τους ε, πολίτες της Ένωσης και για να μπορεί να εφαρμοστεί και η ρήτρα περί προτίμησης των ενωτικών ε, ε, υπαλλήλων. Δεν μιλάμε για μια οδηγία που δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης ή διαφορετικό τρόπο πρόσληψης. Μιλάμε για μια οδηγία που βασίζεται στην νομική βάση της μετανάστευσης και όχι της απασχόλησης. Μιλάμε για τις συνθήκες και τους όρους παραμονής και εργασίας αυτών των ανθρώπων. Παρακαλώ αυτό να το έχετε υπόψη σας όταν διαβάζετε τα άρθρα και όταν σκέφτεσαι πώς θα βελτιωθούν. Ο ορισμός της εταιρεία και του ομίλου. Βεβαίως δεν, είναι δεν υπάρχει ένας ορισμός ενίως και γι' αυτό και στην οδηγία περιλαμβάνεται ένας ορισμός, ώστε τουλάχιστον κάπως να πλαισιωθεί το πράγμα. Και έπειτα θα τα δούμε γιατί δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στο ενοχικό δίκαιο στην Ένωση ώστε να έχουμε έναν ενιαίο ορισμό. Θα πρέπει να δούμε και πώς τα κράτη-μέλη όλα αυτά θα μεταθέσουν, θα μετατρέψουν σε εθνική νομοθεσία. Νομίζω πως θα μπορούσε κανείς να τα δει όλα αυτά από διαφορετική προοπτική, αλλά πάντως το ίδιο, ίδιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στα κράτη-μέλη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ανταγωνίζονται με το εργατικό δυναμικό που ήδη υπάρχει στην Ένωση. Και εκεί που υπάρχει κίνδυνος υπάρχει το τεστ της λειτουργικότητας των διαφόρων επιπέδων και της διαθεσιμότητας τέτοιων ε, ε ανθρώπων ώστε να μην μπορεί κανείς να παρακάμψει τη δυνατότητα να προσλάβει τοπικά, δηλαδή στην Ευρώπη. Βεβαίω μπορούν όλα αυτά να βελτιωθούν, δεν τα αντιλέγω. Αλλά ακριβώς γι' αυτό γίνεται η συζήτηση, ώστε να βρούμε τις απαντήσεις σε, όλα αυτά, σε όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Μπαντάζη τώρα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια και γιατί θέσατε τα συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν και στις συζητήσεις της, ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών ε, φορέων. Πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη ο ορισμοί στην οδηγία για να διευκολυνθεί η εφαρμογή και να υπάρχει ένα διαφανές σύστημα για τους ε, μετατιθέμενους ενδοϊπηρεσιακά και για τις αρχές των κρατών μελών. Έχουμε εντοπίσει αυτή την ανάγκη. Φυσικά σημειώνω και όλα αυτά που είπατε για τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά τα συζητούμε τώρα ενδελεχώς στην ομάδα εργασίας για τα κοινωνικά θέματα. Υπήρξε μια συγκεκριμένη παρατήρηση που θεωρώ ότι πρέπει να την αναφέρω. Η λεγόμενη φυγή εγκεφάλων από τις πιο φτωχές χώρες προς τις πιο πλούσιες. Η οδηγία αυτή νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση υπηρετεί το στόχο του να έχουμε εξειδικευμένους διευθυντές, στελέχη ε, με υψηλή ειδίκευση και πολλά προσόντα για μια μικρή χρονική περίοδο, περιορισμένο χρονικό διάστημα θα παραμένουν. Δηλαδή θα έχουν μια ειδική αποστολή εκτελέσεων και θα επιστρέφουν μετά στις ε, εταιρείε τη χώρα τους. Άρα δεν έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον τον κίνδυνο να υπάρξει διαρροή φυγή εγκεφάλων. Φυσικά η συζήτηση αυτή θα συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς ε, στις αρμόδιες ομάδες του Συμβουλίου και προσβλέπω και εγώ σε όλη τη συζήτηση που θα μας δώσει και μας ε, τροφή και για τις μελλοντικές μας συζητήσεις. Και φυσικά περιμένω να συνεργαστούμε και στο μέλλον στενά με το Κοινοβούλιο αλλά και να ακούσουμε και τους εμπλεκόμενους φορείς. Η κυρία Γιακονσάρη για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πολύ επικοδομητική προσέγγιση. Uh, um, Θα βρούμε λύσεις, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ειδικών εμπειρογνωμών νομίζω ότι πλέον συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι καλό να, να είναι τόσο ευρύς και ευέλικτος ο ορισμός, γιατί τελικά θα υπάρξουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, που θα προσφύγει ο κόσμος στο δικαστήριο. Και αντί να αποφασίσουν οι πολιτικοί θα αποφασίσει το δικαστήριο για το τι εννοούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Μία λύση νομίζω ότι ήδη υπάρχει. Δηλαδή να εμείνουμε αυστηρά στη διατύπωση στο πλαίσιο συμφωνίας GATS, που είναι πιο συγκεκριμένος. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Συμφωνώ επίσης με αυτό το θέμα της φυγής εγκεφάλων. Πράγματι, είναι εύστοχο το ζήτημα που θέτεται. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί θα μπορούσαν να βγουν όλες οι πλευρές κερδισμένες. Δηλαδή τα άτομα αυτά έρχονται στην Ευρώπη και μετά γυρίζουν στην πατρίδα τους και έχουν αποκτήσει ίσως λίγο περισσότερες δεξιότητες από αυτές που είχαν πριν. Όπως και να έχει, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί υπάρχει ένα κοινό πνεύμα. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις και θέλουμε η οδηγία αυτή να είναι στο δυνατόν πιο καλή και ως τον πιο ακριβής και συγκεκριμένη. Διότι δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι τόσο ακριβή όσο θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν με το πρώτο κομμάτι της απογευματινής μας συνεδρίας. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο. Αμέσως θα έλεγα για να προλάβουμε και το χρόνο. Όπως και το πρωί και τώρα έχουμε τρία κομμάτια, τρία σκέλη.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 now leaving for the happy Easter and we welcoming the members of the Καλωσορίζω λοιπόν τους ομιλητές του δεύτερου πάνελ. Οι πρώτοι έφυγαν ήδη για να απολαύσουν το Πάσχα. Good to have you here. Good to have you here. Ecco, ecco, ecco. Ci eh, sbrighiamo subito. We're proceeding, as I said, to the second session. Περνάμε λοιπόν, όπως είπα, στη δεύτερη συνεδρία με συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων. οι οποίοι θα μας μεταφέρουν τις απόψεις τους για την πρόταση της Κομισιόν και για το έργο εργασία του εισηγητή. Έχουμε καλές πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, αλλά και έναν εκπρόσωπο του Eurocadre, που είναι τα στελέχη, επαγγελματικά και διοικητικά στελέχη και φυσικά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πρόταση οδηγίας. Και εν τέλει έχουμε καλέσει και εκπρόσωπο του Ιδρύματος Permits Foundation, Ενό ιδρύματος που έχει ως στόχο την προώθηση της ε, πρόσβαση, της ε, επανένωση των ε, οικογενειών και συγκεκριμένα την εξέβρεση απασχόλησης για τα μέλη της οικογένειας των αποσπασθέντων. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Δίπκε Γάρνεκ, που είναι νομική εμπειρογνώμη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων. Θα σας έλεγα να μιλήσω το καθένα σας πέντε λεπτά για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τους ε, εργαζόμενους ICT, ε, όπως υπόθηκε σήμερα το πρωί και, για σήμερα, και σήμερα το πρωί για την εποχιακή εργασία, έχουμε κάποια προβλήματα και έχουμε και κάποιες λεπτομερείς παρατηρήσεις όσον αφορά την πρόταση για τους ε, εσωτερικά αποσπαστέντες, τους ICT. Υπάρχει μια τάση ε, κατάκμησης της αγοράς εργασίας, όπως ανέφεραν σήμερα το πρωί οι συναδελφοί μου και δημιουργούνται διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Για μας λοιπόν αυτή είναι μια πρόταση που υποθάλπει τον αθέμητο ανταγωνισμό, υπονομεύει την ίση μεταχείριση, ε, την αρχή της ε, χώρας ε, και την διαπραγματευτική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Γι' αυτό λοιπόν τα αιτήματά μας ε, με βάση την πρόταση είναι τα εξής και θα μπω ε, σε λεπτομέρειες μόνο στο βασικό μας αίτημα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι θα θέλαμε να υπάρχει μια διπλή νομική βάση. Βεβαίως συμφωνούμε ότι η νομική βάση στη μετανάτευση είναι σωστή, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει, να προσθεθεί και άλλη μία νομική βάση. Φαντάζομαι δεν θα αρνηθείτε ότι η οδηγία αυτή θα επηρεάσει την αγορά εργασίας. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για ένα εργαλείο ε, το οποίο ορίζει την είσοδο και την εγκατάσταση, τη διαβίωση ε, των μεταναστών εργαζομένων. Ε, πρόκειται και για τον ορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων αυτών. Και ομολογώ εξεπλάγην που προηγουμένως ε, στο πάνελ δεν μιλήσαμε τόσο για τους εργαζόμενους όσο για τις εταιρείες τους. Βασικά μας αιτήματα είναι λοιπόν η ίση μεταχείριση και η μη διακρίση. Άρθρο 14 των δικαιωμάτων, αυτό μας απασχολεί κατά κύριο λόγο. Και βλέπουμε εδώ να υπάρχουν δύο προβλήματα σε αυτό το άρθρο. Το ένα είναι ότι οι ασυτείς αντιμετωπίζονται ως αποσπαστέντες εργαζόμενοι που ε, σημαίνει ότι αν τελικά προσπίβεται ότι υπάρχει ίση μεταχείριση στην οδηγία ναι, ας το δεχτούμε, αλλά με μια κατηγορία εργαζομένων, των αποσπασμένων, οι οποίοι ήδη έχουν ελάχιστη ε, προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόφαση του ΔΕΚ. Και γνωρίζουμε ότι ε, δεν θα υπάρξει καμία σχετική διάταξη, δεν θα προσθεθεί καμία διάταξη σε αυτήν την οδηγία. Το δεύτερο πρόβλημά μας είναι η παραπομπή σε συλλογικές συμβάσεις με ευρεία εφαρμογή ε, και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ είναι απαραίτητο να υπάρξουν διαγραφές διαγράψουμε κάποια κομμάτια της οδηγίας. Γιατί επιθυμούμε οι εργαζόμενοι αυτοί, οι ICT, να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλα τα επίπεδα των συλλογικών συμβάσεων. Άρα δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι τα κριτήρια εισόδου των εργαζομένων. Εκεί οι 12 μήνες απασχόλησης ε, πριν από την απόσπαση για μας ε, είναι σημαντικό αυτό να είναι υποχρέωση ε, των κρατών μελών και όχι επιλογή τους. Και χάρηκα πάρα πολύ που αυτό το θέμα το ανέφερε και ο εισηγητής. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε αναμφισβήτητα τους 12 ε, μήνες ε, για να έχουμε ε, μία πραγματική σχέση. Και όπως ακούσαμε και προηγουμένως, έχουμε προβλήματα με τον ορισμό, κυρίως τον ορισμό ε, των εξειδικευμένων και των μάνατζερ. Τέλος πάντων, το θέμα αυτό θα τεθεί από τους συναδέλφους από την EuroCard, αλλά θεωρούμε απαραίτητα ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός του ορισμού. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι πολύ ευρύ ε, και εξεπλάγει που ο κύριος Μανσαβίζη ανέφερε ότι εδώ πρόκειται για μια οδηγία που αφορά στις ε, πολυεθνικές. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται στην οδηγία ότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το είδος και το μέγεθος της εταιρεία και όχι στους κλάδους. Θα γνωρίζετε ενδεχομένως ότι ο τομέας των κατασκευών ζητήθηκε να εξαιρείται από αυτή την οδηγία γιατί φοβούνται ότι η οδηγία αυτή δεν θα βοηθήσει τον τομέα. Ε, και αυτή είναι μια εξαίρεση την οποία δέχτηκαν και οι κοινωνικοί εταίροι. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να πω ε, είναι ότι δεν υπάρχουν, λείπουν ε, αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου. Όσον αφορά το έγγραφο εργασία ε, του κ. Διακολίνο, μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με πολλά από αυτά που αναφέρει, αλλά δεν υπάρχουν για μας δύο βασικά αιτήματα που, όπως σας είπα, είναι τα δικαιώματα των ITC εργαζομένων το, ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και λείπει και η σύνδεση με την οδηγία περί αποσπάσεων. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο για δεύτερη φορά σήμερα στον κύριο Ρούντεμπεργκ, τον οποίο καλωσορίζω για δεύτερη φορά. Πρόκειται για τον πρόεδρο τη Ομάδα Εργασία σχετικά με τη μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για τη Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, το Business Europe. Έχετε το λόγο, κύριε Ρούντεμπεργκ. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ σωστά. Εκπροσωπώ την Business Europe, που είναι η εταίρη σας από τη Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, δηλαδή εκπροσωπούμε τις οργανώσεις επιχειρηματιών και εργοδοτών από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εκπροσωπούμε ευρωπαϊκές εταιρείες. Και θα επανέλθω σε αυτό όταν μιλήσω για την ε, μετάθεση υπαλλήλων εκτός Ευρώπης. Νομίζω όμως ότι υπάρχει κάποια σύγχυση για το τι ακριβώς είναι αυτή η οδηγία και τι είναι και τα EICTs ή υπηρεσιακός μετατιθέμενοι. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την κινητικότητα εργαζομένων με υψηλή δίκευση, οι οποίοι έχουν ήδη συμβόλαιο σύμβαση απασχόληση και διατηρείται αυτή η σύμβαση όταν αυτοί οι υπάλληλοι μετατίθενται από έναν φορέα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εταιρεία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρούν και την απασχόλησή του, τη θέση του. και είναι πολύ σωστό το ότι επιλέγει να πει η Κομισιόν ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για την οδηγία, ε, της οδηγίας περί απόσπασης, διότι υπάρχει μια ομοιότητα Ήδη δηλαδή ο υπάλληλο έχει μία θέση εργασία, τη διατηρεί και μετά τη μετάθεσή του. Βέβαια η απόσπαση, η οδηγία περί απόσπασης δεν ισχύει γιατί η εταιρεία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να μην παρέχει απαραίτητος υπηρεσίες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστή η προσέγγιση της Κομισιόν. Εάν λοιπόν έχουμε αυτούς τους κανόνες για τα δικαιώματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αποσπασθέντες εργαζόμενους, νομίζω ότι αυτό επαρκεί και είναι κατάλληλο όταν μιλάμε για την μετάθεση ε, υπαλλήλων από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μεταθέτει ενδοϊπηρεσιακά ξέρουμε ότι είναι βαθμό στέλεχη ό,τι αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και τα άτομα αυτά μπορούν να διαφυλάξουν και να προσπίσουν τα συμφέροντά τους με πολύ καλό τρόπο. Δηλαδή αν δεν ε, θεωρούν ότι οι συνθήκες και οι όροι είναι ικανοποιητικοί δεν πρόκειται πολύ απλά να φύγουν από τη χώρα τους και να πάνε σε μια άλλη. Οι εταιρείε δεν μεταθέτουν αυτά τα άτομα τους ICTs γιατί είναι φθηνό εργατικό δυναμικό. Όχι, γιατί είναι δαπανηρή η μετάθεση ενός ε, υπαλλήλου από τη μια χώρα στην άλλη. Μετακίνηση, στέγαση και όλα τα άλλα που συνδέονται. Γίνεται αυτό από τις εταιρείε γιατί είναι απαραίτητο, γιατί είναι καλό και γιατί ε, μπορούν να το κάνουν πράξη λόγω της οργάνωσης που έχουν. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, ανεξαρτήτως του πόσο ορίζεται στην οδηγία, μιλάμε εδώ για ειδικέ γνώσεις. Δεν μιλάμε για την ε, παιδεία, την εκπαίδευση που έχει το άτομο, αλλά μιλάμε για ειδικέ γνώσεις ε, ε, αγοροκεντρικές ή προσανατολισμένες στο προϊόν. Δηλαδή, έχει το άτομο αυτό, αυτές τις γνώσεις που έχει ως αποτέλεσμα να η καλύτερη λύση είναι να το μεταθέσει σε μια άλλη χώρα στην εταιρεία. Επαναλαμβάνω ότι είναι δαπανηρή λύση, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά για μια προσωρινή επαναλαμβάνουμε αποστολή. Σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφος από τα συνδικάτα, η λέξη πολυεθνική multinational δεν χρησιμοποιείται στην οδηγία. Μιλάμε για την απόσπαση ενός εργαζομένου ο οποίο μεταφέρεται από ένα φορέα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν άλλο φορέα εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε τελικά για πολυεθνική, κατά την άποψή μου, για πολυεθνικέ εταιρείε. Τίνουμε να συζητήσουμε τώρα το αν είναι α, Ινδική, Αμερικανική ή Ευρωπαϊκή εταιρεία. Η ταυτότητα της εταιρεία ό,τι αφορά όμως ε, την εθνικότητα δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ευρωπαϊκές εταιρείε οι οποίες έχουν κάποια ε, παραρτήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η IBM ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που αντιστρόφως στέλνει ε, υπαλλήλους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα, παραλαμβάνω, δεν είναι η, η εθνικότητα, αλλά οι γνώσεις. Οι γνώσεις είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και εμείς ως εκπρόσωποι εταιρεών από την Ευρώπη θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Το να μπορούμε δηλαδή να μεταφέρουμε δεξιότητες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστό είναι αυτό που λέγεται ότι είναι δύσκολο να δει κανείς πώς αυτό θα επηρεάσει τον αριθμό των ατόμων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νούμερα. Δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ίσως Τώρα, αν θα αυξηθούν τα νούμερα δεν ξέρουμε, αλλά είναι δυνατό πλέον να μεταφέρεται ένα άτομο από το ένα κράτος στο άλλο, αφού το άτομο αυτό μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προτείνεται στην οδηγία. Εναρμόνιση και επιτάχυνση διαδικασιών, αλλά και ενδοκινοτική κινητικότητα. Και εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για προτάσεις νομικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενδοκοινοτική, η ενδοενωσιακή πτυχή είναι ο λόγος ύπαρξης, που αυτό είναι που θα δώσει προστιθέμενη αξία. Είναι ένα θέμα λεπτό που αφορά την κυριαρχία των εθνικών κρατών μελών, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πιστεύω δε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Είδαμε τι έγινε και με την κρίση την πρόσφατη, αν αυτός ο παράγοντας δεν συντρέχει. Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα και συγκεκριμένα την τελευταία μου διαφάνεια, επειδή δεν έχω χρόνο, σας αφήνω να τη διαβάσετε μόνοι σας. Οπότε θα έχετε έτσι σχηματίσει μία πλήρη άποψη και θα έχετε και το πλήρες έγγραφο εργασίας της Business Europe. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μπορώ να σας πω ότι αργότερα στην τρίτη συζήτηση θα ακούσετε από τον κύριο Κόξ και από, ε, από τους κύριους Κόξ και Νιψάρ πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα και γι' αυτό παραμείνετε σας παρακαλώ εδώ για να ακούσετε και τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούντε Μπέρκα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ξέραμε ότι έχετε τις διαφάνειες. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Μισελ Πατάχ, αντιπρόεδρο του Eurocadre. Έχετε το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την Επιτροπή για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Για να σας παρουσιάσω την Eurocadre, είναι μια, ε, ένα σύνδεσμος αναγνωρισμένος, ενεργός και, και συγκεντρώνει 6 εκατομμύρια στελέχη με ένα επίπεδο εκπαίδευση ευθυνών και αυτονομίας πολύ σημαντικό και είναι αναπόσπαστο τμήμα της, ε, του πληθυσμού τον οποίο στοχεύει αυτή εδώ η πρόταση. Η Eurocadre είναι βασικά υπέρ τη κινητικότητα, της κινητικότητα του προσωπικού, του υψηλά ειδικευμένου μάλιστα, πράγμα το οποίο αυξάνει και την ε, κινητικότητα των γνώσεων και του ταλέντου και αυξάνει και τις δυνατότητες αδιοδρομίας για τα στελέχη. Θεωρούμε επίσης ότι οι στόχοι αυτής της οδηγίας, της πρώτας οδηγίας είναι σωστοί, δηλαδή να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να μπορούν να μετακινούνται οι προσοντούχοι υπάλληλοι που είναι τουλάχιστον προσωρινά απαραίτητοι σε άλλες έδρες εταιρεία. Ωστόσο, από την άποψη των στελεχών στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής ώστε αυτή να καταστεί πιο λειτουργική για τα στελέχη και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Πριν να έρθω στην μορφή της, ε, της οδηγίας, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί της ουσίας. Καταρχήν, τα μέλη του Eurocadre γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μέγα αριθμό τελεχών θα φύγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια και ότι δυστυχώς ο αριθμό των νέων διπλωματούχων στην Ευρώπη δεν θα αρκέσει ιδιαίτερα για να αντικατασταθούν οι γενναίες που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1950 και το 1965. Άρα λοιπόν αυτή η οδηγία είναι και καλύπτει μια νέα πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως η συζήτηση γίνεται σε μια πολύ άσχημη συγκυρία με την κρίση που ταλανίζει, την κοινωνική κρίση που ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι είναι συχνά θύματα γιατί δεν βρίσκουν εύκολα σταθερή δουλειά, είτε το δίπλωμά τους, το πτυχίο τους υποτιμάται. Ε, ε, όσον αφορά την πρόσληψή του, μάλλον κατά την πρόσληψή του. Άρα λοιπόν η εφαρμογή αυτή τη οδηγία θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά εργασία στην Ευρώπη και η Eurocadre θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των διπλωματούχων είτε είναι ε, πολίτε Ένωση είτε όχι. Α έρθουμε τώρα στην μορφή. Η Eurocadre συμμερίζεται το σχέδιο γνωμοδότης που θα επευληθεί σε έγκριση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στι 4 και 5 Μαου. Ε, δεν επανέρχομαι στο θέμα που συνδέεται με την ισότητα ε, μεταχείρισης. Ήδη αναφέρθηκε η συνάδελφος από την ETUC, ούτε και στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που για την ε, Eurocat χρειάζεται νέα σύνταξη. Θα μιλήσω για τα προβλήματα που τίθενται λόγω της οριστείας ορισμένων ορισμών και ιδιαίτερα όσον αφορά τους ορισμούς E, F και Z του άρθρου 3, δηλαδή τον πληθυσμό που θα ε, διέπεται από αυτές τις διατάξεις. Ε, καταρχήν ε, για τους μάνατζερ λέτε, μάλλον μιλάτε για τα διοικητικά στελέχη, αλλά ο, ο, ορισμός τελικά αναφέρεται σε όλα τα στελέχη που εποπτεύουν την εργασία και που έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν ή να απολύσουν άλλο προσωπικό. Και αυτό ξεπερνά τους μάνατζερ και διευρύνεται στην μεγάλη μάζα των όσων οι Γάλλοι αποκαλούν τα στελέχη των στελεχών, τα που στελεχώνουν τα στελέχη ή που πλαισιώνουν τα στελέχη. Ε, τώρα, όσον αφορά τους ειδικού, η Eurocat πιστεύει ότι αυτός ο ορισμός μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο του ειδικευμένου εργαζόμενου, αλλά και του περισσότερου τεχνικού, από τη στιγμή που έχουν ένα επίπεδο πτυχίου που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο ανώτατη εκπαίδευση. Αυτός ο ορισμός λοιπόν ως έχει μπορεί να επιτρέψει την μετακίνηση ενός σημαντικού αριθμού υπαλλήλων μια εταιρεία, που δεν νομίζουμε ότι αντιστοιχεί στον πληθυσμό που θέλει να καλύψει η οδηγία. Ε, και από αυτού θεωρούμε ότι η σημερινή ακρόαση θα επιτρέψουν να διευκρινιστούν οι ορισμοί αυτοί. Όσον αφορά τώρα τους σταζιέρ, ή υποδοκιμοί και εκπαιδευόμενους ή υπό δοκιμή. Και εκεί είναι μεγάλο, μεγάλη οριστια γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές για τον ορισμό αυτών των ανθρώπων στις χώρες μέλη της Ένωσης ε, ένα σταζιέρ μπορεί να είναι είτε πτυχιούχος που τελειοποιείται ε, μέσω μιας ειδίκευσης σε μια εταιρεία είτε αντίθετα μπορεί να είναι ένας ε, φοιτητής ο οποίος προετοιμάζει την πτυχιακή του εργασία και που η δουλειά του σε αυτή την επιχείρηση θα χρησιμεύσει ως ε, προϋπηρεσία και προαπαιτούμενο για την το πτυχίο του. Επίσης οι συνθήκες αμοιβή είναι πολύ διαφορετικές. Το να συμπεριληφθούν λοιπόν οι ειδικευόμενοι, ακόμα και αν προετοιμάζονται για να γίνουν ανώτατα στελέχη, θα ήταν ε, νομίζω υπερβολικό. Θα έπρεπε να υπάρξει ένα τελείως διαφορετικό ε, καθεστώς που θα έμοιαζε ίσως με το πρόγραμμα Εράσμους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, τώρα... Ναι, τα πήγατε πολύ καλά. Με το χρόνο έχουμε πάει πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν έχουμε την κυρία Κάθριν Βαντεουίλκ που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πέρμιτς. για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμβάλλω και εγώ στη συζήτησή σας ε, για τις ε, ενδοεπιχειρησιακές ε, αποσπάσεις. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στα μέλη των οικογενειών, δηλαδή στην πρόσβασή τους στην απασχόληση και επίση και στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να έχει διεκπαιρεωθεί η αίτησή τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή που αναφέρεται και στα δύο θέματα στο έγγραφο εργασίας που συνέταξε για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Η δική μας οργάνωση, η Permits, το Ίδρυμα Permits, είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμός που προάγει την δυνατότητα απασχόλησης ε, ε, μελών οικογενειών. Ε, έχουμε 40 εταιρείε, σημαντικέ εταιρείε που είναι χορηγοί μα. και ο αριθμός των εργαζομένων που έχουμε βοηθήσει να βρουν εργασία είναι περίπου πάνω από 2 εκατομμύρια. Βεβαίως, μιλάμε για το 1% του συνόλου των απασχολωμένων. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, αν λάβει κανείς ε, υπόψη του ότι οι άνθρωποι αυτοί διευκολύνουν κατά πολύ και ενισχύουν κατά πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς χαιρετίζουμε τις προτάσεις της Επιτροπής και στηρίζουμε αυτά τα οποία ανέφερε κυρίως η Business Europe. Εμείς επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε ότι όσον αφορά την πολιτική για το προσωπικό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη της οικογένειας στο σύνολό της. Ε, σήμερα Υπάρχουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά την απασχόληση του ή της συντρόφου και αυτό είναι βασικός λόγος γιατί κανείς απορρίπτει μία προσφορά εργασίας. Εμείς λοιπόν ως Ίδρυμα ε, σας καλούμε να προτείνετε δύο τροπολογίες στο άρθρο 15. Πρώτον, θα θέλαμε να υπάρχει μια νέα ρήτρα που θα επιτρέπει ε, στα συνοδά μέλη οικογενειών να βρουν άμεσα θέση απασχόλησης. Κάτι το οποίο συμβαδίζει με την διατύπωση που ε, υπάρχει στην οδηγία περί μπλε κάρτας. Δεύτερον, τα μέλη των οικολογιών, οικογενειών ε, θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής ε, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα των 30 ημερών και όχι σε δύο μήνες όπως αναφέρεται στην οδηγία ε, μερικές φορές ίσως βολεύει να έρθουν οι σύντροφοι αργότερα για να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο αλλά κατά κανόνα είναι φυσιολογικό να έρθει όλη η οικογένεια μαζί. Είναι επίσης σημαντικό ε, το ότι ε, ορισμένοι από τους αποσπαζόμενους προέρχονται από άλλη χώρα που είχαν πάλι αποσπαστεί ένας Αμερικανός ας πούμε ε, που έρχεται στην Ευρώπη μπορεί να έρχεται από το Χονγκ Κόνγκ ή από το Ντουμπάι και από τη στιγμή που ο εργαζόμενος φεύγει από την χώρα στην οποία ήταν επίσης εκπατρισμένος η οικογένεια πρέπει να έχει το δικαίωμα να παραμείνει εκεί ε, και όταν έρχονται στην Ευρώπη επίσης να μπορούν να έρχονται όλοι μαζί. Όσον αφορά τώρα το θέμα της πρόσβασης στην απασχόληση των συντρόφων ε, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή περίπου 20 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο επιτρέπουν στις ε, συνοδούς ε, γυναίκες, συζύγους και παιδιά να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό αφορά 11 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν η Ένωση στο σύνολό της ε, δεν συμβαδίσει με την βέλτιστη πρακτική σε διεθνές επίπεδο θα χάσει πολύτιμα ταλέντα και θα αποδυναμωθεί οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από το πρίσμα των ίσων ευκαιριών ε, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το 85% των συνοδών συντρόφων είναι γυναίκες που σημαίνει ότι όταν δεν δίνεται άδεια εργασία και στους δύο συντρόφους, αυτό ε, πλήττει κατά κύριο λόγο τις ε, γυναίκες ε, και οι γυναίκες πολλές φορές δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν και πρόσβαση σε κρατικούς πόρους. Αυτό όμως δεν είναι ίση μεταχείριση, κάτι το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 79 Τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί προβλέπεται η συμμεταχείριση για όλου όσοι διαμένουν στην Ευρώπη. Αντίθετα, τον επιτρέψει κανεί στου συντρόφου να εργαστούν κατά τη διάρκεια ενό συγκεκριμένου συμβολέου, αυτό σημαίνει ότι μπορούν και οι ίδιοι να διατηρήσουν τα προσόντα του και όταν επανέλθουν στην πατρίδα του να ενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασία. Αυτό συμβάλλει στην κυκλική μετανάστευση και βελτιώνει τι προοπτικέ απασχόληση και στη χώρα αποστολή και στη χώρα προέλευση. Το Ίδρυμα Permits έχει και περαιτέρω στοιχεία από μία έρευνα που κάναμε σε 3.000 ε, συζύγου και συντρόφους, ε, συνοδού ε, αποσπασμένων εργαζομένων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αποδείχτηκε ότι ε, ένα τέταρτο προσωπικού εργαζομένου σε διεθνές επίπεδο απέρριψαν προσφορά λόγω της καριέρας ε, της συντρόφου ή του συντρόφου και περίπου το 60% είπαν ότι στο μέλλον δεν θα μεταβούν σε χώρα όπου θα είναι δύσκολο για τον σύντροφο να βρει εργασία. Βλέπετε λοιπόν τι πρόκληση υπάρχει ε, όταν, λέμε, όταν μιλάμε για την προσέλκυση των άριστον και αυτά θα χειροτρέψουν ακόμα περισσότερο λόγω της δημογραφικής αλλαγής. Εξάλλου, μέσα στην έρευνα πολλές γυναίκες είπαν ότι όσες είχαν εργασία είχαν καλύτερη προσαρμογή, καλύτερες οικογενειακές σχέσεις, καλύτερη υγεία και ευημερία. Πολλές γυναίκες έκαναν και άλλα σχόλια ε, και θα ήθελα να φέρω ένα από εσάς φτάνοντας στο συμπέρασμά μου. Ε, μία γυναίκα από μη κοινοτική χώρα ε, που συνοδεύει το σύζυγό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από πολλά χρόνια που εργάστηκε είπε και παραθέτω τώρα που επανέρχομαι στο χώρο της εργασίας θα είναι ψυχολογικά πολύ δύσκολο να κάνω και πάλι διακοπή, διάλειμμα ή να ε, σε άλλη χώρα. Έχει τεράστια διαφορά στο πώς με αντιμετωπίζουν τα παιδιά μου. Ε, τα παιδιά μου με αντιμετώπιζαν ως μητέρα, ως σύζυγο και τώρα με αντιμετωπίζουν ως επαγγελματία. Και αυτό επηρεάζει και τις δικές τους τι προσδοκίες. Ε, τα σχόλια της ε, κόρης μου ήταν... Ε, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι και τα, και τα κορίτσια μπορούν να εργάζονται και να είναι και μητέρες. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα ξεπερνάει τις ε, άμεσες ε, επιπτώσεις από τη διαδικασία αυτή επιλογής των άριστον. Το Ίδρυμα Permits πιστεύει ότι πραγματικά εδώ υπάρχει μια ευκαιρία ε, να προκύψει τριπλό όφελος, δηλαδή για τις οικογένειες, για τις εταιρείε, αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να ε, εγκρίνετε τις απαραίτητες τροπολογίες στο άρθρο 15 και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα θελήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φαντεμβίλκ. Ώρα για συζήτηση. Θέλει κάποιος από τους συναδέλφους το λόγο. Κανείς. Δεν έχετε ερωτήσεις. Αν δεν έχετε ερωτήσεις δεν υπάρχει και απάντηση. Άρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Α, η κυρία Μορβάη. Μια σύντομη παρατήρηση ανακούφισης ε, που σημαίνει επιτέλους μιλάμε για υψηλό για υψηλές, και υψηλά στελέχη με πολλά προσόντα. Τι ανακούφιση που το 85% είναι άντρες. Ναι, πράγματι. Ήταν ακριβώς ένα σχόλιο που είχε να κάνει ακριβώς με αυτά που λέγατε. Κύριε Μούλτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έθεσα το ίδιο ερώτημα και στον προηγούμενο γύρο. Τι γίνεται σε ΣΥΠΑ, στην Ινδία, στην Κίνα. Υπάρχουν αντίστοιχε νομοθεσίες ε, σε άλλου εμπορικού μα εταίρου η κυρία Φάντερ Βίλκ. Εμεί στο πλαίσιο τη διεθνού μα έρευνα έχουμε μετρήσει, έχουμε μάλλον μελετήσει πάνω από 20 χώρε θα μπορούσα να σας πω κάποια στοιχεία. Στην Ευρώπη, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες έχουν εγκρίνει κάποια νομοθεσία. Οκτώ συνολικά χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σύντροφος ή οι σύντροφες μπορούν να εργαστούν. Η Γερμανία, εργαστουν γερμανια βελγιο και Ιρλανδία τώρα, αν υπάρχει προσφορά για θέση εργασίας, δίνεται και άδεια εργασίας και στο σύντροφο. Αυστραλία, Ελβετία, ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία κτλ. Υπάρχει και σε, και σε κάποιες άλλες χώρες, στο Μεξικό, τη Σιγκαπούρη, υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις. Γενικώ αυξάνονται οι χώρες γιατί επειδή επεκτείνεται αυτή η πρακτική έχουν αντιληφθεί και οι εργοδότες τη σημασία που έχει ο σύντροφος να συνοδεύει και να εργα... τον ε, σύντροφο και να εργάζεται. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίως το θέμα της αμοιβαιότητας. Όταν ε, μιλάμε ε, για τις ε, ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχουν οι πολυεθνικές να μεταθέσουν τους υπαλλήλους Γνωρίζουμε όλοι ότι γίνονται διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο ε, της συμφωνίας GATS, αλλά υπάρχουν και διμερείς ε, συμφωνίες και τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη διαπραγματευτική θέση όσον αφορά στην αμοιβαιότητα. Να μπορεί κανείς δηλαδή να μεταθέτει υπαλλήλου και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται όλα αυτόματα, αλλά νομίζω ότι κάνουμε το σωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πρωτοπόροι ε, και νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα ε, καλύτερα αποτελέσματα. Ο συνάδελφός μας από τη Γαλλία ε, θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, να επανέλθω σε μια συζήτηση που έγινε και στην προηγούμενο πάνελ όσον αφορά τη φυγή των εγκεφάλων. Νομίζω ότι για το θέμα των πτυχιούχων είμαστε περίπου στο ίδιο, στην ίδια κατάσταση όπως και για τους εποχικούς εργαζόμενους σήμερα το πρωί. Επειδή έχω συζητήσει με τα Σενεγαλέζικα Συνδικάτα τον Ιανουάριο, πάνω από το ίμιση των μεταναστών από τη Σενεγάλη είναι νέοι πτυχιούχοι οι οποίοι δοκιμάζουν την τύχη τους ιδιαίτερα στην Ευρώπη και όχι απαραίτητο στις ε, θέσεις ε, όπου απαιτούνται πτυχία, αλλά πολύ συχνά σε θέσεις ε, που με πολύ χαμηλούς μισθούς. Και σήμερα το πρωί αναφέρθηκε και η Ουγγαρία και η Εκτελεστική Επιτροπή της Eurocountry ήταν στην Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα και φαίνεται πως οι νέοι Ούγγροι διπλωμα... πτυχιούχοι προσπαθούν καταρχήν να βρουν δουλειά σε επιχειρήσεις στην Αυστρία και στην Πολωνία Πολωνία. Δηλαδή αυτό το θέμα της φυγής εγκεφάλων υπάρχει σήμερα. Μα υπάρχει στο βαθμό που το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων και των δεξιοτήτων των προσόντων και βία αυτών τίθεται Τίθεται ούτως ή άλλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά με την εξέλιξη των ανταλλαγών σε πλανητικό επίπεδο, τίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει ο συνδικαλισμός, ε, ιδιαίτερα ο συνδικαλισμός που αντιπροσωπεύει τα στελέχη να δουλέψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν πραγματικά να έχουν ε, συνθήκες δουλειάς και αμοιβή στη χώρα τους ε, επαρκής και να μπορούν να μείνουν στη χώρα τους. Είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο δουλεύουμε με τα αφρικανικά συνδικάτα, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση των πτυχιούχων στην Αφρική είναι καταστροφική. Ευχαριστώ. Merci à Ευχαριστώ κύριε Πατέρα. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ. Γιατί έχουμε ακόμα ένα πάνελ. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ομιλητές μας σε αυτή τη δεύτερη συνεδρία και πάμε για τον τρίτο γύρο.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 Ε, σας ευχαριστούμε που έχετε την καλοσύνη να μας ε, βοηθήσετε να ε, τελειώσουμε στην ώρα μας σήμερα το απόγευμα. Πολλοί από εμά περιμένουν να πάνε διακοπές για το Πάσχα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να μπουν στα αεροπλάνα, να πετάξουν, να σεβαστούμε το ωράριο. Με αυτό λοιπόν στο μυαλό μας πάμε στο τρίτο τμήμα του σημερινού απογεύματος που αφορά πρακτικά παραδείγματα. Τώρα λοιπόν θα ασχοληθούμε με πρακτικά παραδείγματα ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων και αποφασίσαμε να ε, καλέσουμε εκπροσώπους δύο επιχειρήσεων που συνδυάζουν και συσχετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολυεθνικές. Ε, είναι Ινδικές ε, πολυεθνικές εταιρείε που έχουν παρουσία στην Ινδία, η πρώτη περίπτωση, Ευρωπαϊκό Αμερικανικό Business Council. Θα ακούσουμε τη δική τους άποψη για την ε, πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ακούσουμε λοιπόν την άποψή τους και ε, θα προβλέψουμε και κάποιο χρόνο για συζήτηση πριν ακούσουμε την ανακεφαλαίωση από τον κύριο Γιακολίνο, τον εισηγητή μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καρλ Κόξ, που τον χαιρετίζουμε θερμά. Είναι συμπρόεδρος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, Εξειδικευμένων Εργαζομένων. Κύριε Κόξ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω και κάποιες διαφάνειες που θα συνοδεύσουν τις εισηγωγικές μου παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε και εσείς, ε, εκπροσωπώ το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Επιχειρήσεων, ε, που είναι ο μεγαλύτερος περατλαντικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και στην Ευρώπη, λοιπόν, και στις ΗΠΑ έχουμε 72 εταιρείες μέλη που ουσιαστικά εκπροσωπούν όλους τους τομείς παγκόσμιας οικονομίας, φαρμακοβιομηχανία, τεχνολογίες των πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες, ε, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορία, συμβουλευτική, καταναλωτικά αγαθά. Εμείς χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη διευκόλυνση της εισόδου των ε, ενδοϊπηρεσιακά μετατεθεμένων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν νωρίτερα, η σχετική οδηγία αντικατοπτρίζει το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο που μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ε, ανάγκες σε δεξιότητες και ε, ταυτόχρονα ε, ελατω, ελαττωμένα ποσοστά εξειδικευμένων αποφύτων πανεπιστημίων σε διάφορους τομείς σε διάφορα αντικείμενα. Και επομένως εμείς ανησυχούμε, ανησυχούμε όλο και περισσότερο και δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να βρούμε άτομα με υψηλή εξειδίκευση τα οποία θα είναι διαθέσιμα να πάσα ώρα και στιγμή και σε κάθε αγορά όταν τους χρειάζονται οι πελάτες μας. Έτσι λοιπόν αυτή η οδηγία η οποία και επιτρέπει και διευκολύνει τη δυνατότητά μας να φέρουμε ειδικευμένου υπαλλήλου και τις δεξιότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινό χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μου ζητήθηκε συγκεκριμένα να ασχοληθώ με τις πρακτικές ε, πτυχές αυτής της εδώ υπηρεσιακής μετάθεσης. Ε, δηλαδή πότε επιλέγει ένας εργοδότης να φέρει έναν ειδικευμένο υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα. Δύο παραδείγματα, δύο πιθανά σενάρια ε, θα ήθελα να σας περιγράψω. Φυσικά υπάρχουν πολλά διαφορετικά παραδείγματα, πολλά διαφορετικά σενάρια. Δύο όμως θεωρώ άξια συζήτηση εδώ. Ας πούμε ότι ένας πολιτής ε, λογιστικού από τις ΕΠΑ εγκαθιστά ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού σε μια ισπανική εταιρεία ή εφαρμογή του λογισμικού θα επιταχύνει την παράδοση των υλικών στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα μειώσει την ανάγκη απογραφής και θα έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολύ μεγάλες οικονομίες για την ισπανική αυτή εταιρεία. Πριν όμως ε, ξεκινήσει η ανάπτυξη αυτού του λογιστικού υπάρχει ένα πρόβλημα, ανακύπτει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να ξεκινήσει η δοκιμή αυτή τη εφαρμογή εάν δεν λυθούν τα προβλήματα. Επειδή αναπτύχθηκε αυτή η εφαρμογή στη ΣΥΠΑ, εκεί υπάρχει και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουν μηχανικοί, μηχανολόγοι λογισμικού, το συντομότερο δυνατό, για να λύσουν ε, προβλήματα στις αποθήκες του, ε, του πελάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραμείνουν επιτόπου για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα προκύψουν άλλα προβλήματα και πριν αλλά και μετά την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής. Αυτό είναι ένα σενάριο και θα επανέλθω αργότερα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με μια μεγάλη μεταποιητική εταιρεία από την Γερμανία όχι με έδρα ε, εκτός Ένωσης, με έδρα εντός Ένωσης. Αυτή η εταιρεία πρόσφατα προσέλαβε ελπιδοφόρα νεαρά στελέχη από πέντε ταχιώς αναπτυσσόμενες χώρες, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Αυτοί οι πήκοοι τρίτων χωρών έρχονται στην έδρα ε, της εταιρείας στη Γερμανία για έξι μήνες ε, προκειμένου να ε, συμπήξουν σχέσεις με τη, τα διευθυντικά στελέχη, να μάθουν τις εσωτερικές διεργασίες, διαδικασίες, αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και αναδυόμενες αγορές για τις οποίες ε, είναι υπεύθυνοι και για να κατανοήσουν καλύτερα ε, τα διάφορα ε, προγράμματα και τις διάφορες στρατηγικές κατευθύνσεις. Και μετά θα επανέλθουν στη χώρα τους και θα εργαστούν σε ηγετικές θέσεις στις θηγατρικές της γερμανικής αυτής εταιρείας. Η οδηγία λοιπόν ICT μπορεί να διευκολύνει τέτοιε περιπτώσει σαν που σα εξέθεσα ως παραδείγματα και οι επιχειρήσεις αυτές να μπορούν έτσι να έχουν τα καλύτερα ταλέντα στη διάθεσή τους, να μπορούν να τα φέρουν από ολόκληρο τον κόσμο σε επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πελάτες μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αρκετή αναφορά της αξίας που μπορεί να φέρουν αυτοί οι μετατιθέμενοι πάλι όχι μόνο στους εργοδότες του, αλλά στους πελάτες. Αυτό νομίζω δεν έχει τονιστεί αρκετά γιατί, παραδείγματος χάρη, ε, στο πρώτο παράδειγμα θα εργάζονται για μια ισπανική εταιρεία αγαθών, εμπορευμάτων, άρα δεν εργάζονται μόνο προς όφελος των εργοδοτών αλλά και προς όφελος των πελατών στην Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας λοιπόν υπάρχουν κάποιες βασικές πτυχές της πρόταση που είναι σημαντικέ για τις επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω ούτε μπορώ να δούμε ε, τώρα αναλυτικά για τις 13 αυτές ε, πτυχές. Απλά θα ήθελα σε πέντε από αυτές να εστιάσω προτού ολοκληρώσω. Στα δύο παραδείγματα που σας εξέθεσα σε ό,τι αφορά την εταιρεία λογισμικού από τη ΣΥΠΑ και τη γερμανική μεταποιητική εταιρεία. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία Πρώτα απ' όλα οι διατάξεις ενδοενασιακής κινητικότητας. Σας είπα για την ε, Αμερικανική Εταιρεία Λογισμικού και την Ισπανική Εταιρεία που έχει αποθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα αυτός ο υπάλληλος που μετατέθηκε δεν εργαζόταν μόνο στην Ισπανία, θα έπρεπε να πάει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, ο υπάλληλο αυτός, ο μετατιθέμενος, θα πρέπει να εργάζεται όχι μόνο σε καταστάσει ε, του εργοδότη, αλλά και σε καταστάσει των πελατών. Όπω ε, είναι σαφέ και από το παράδειγμα, παραδείγματο χάρη αυτοί οι μηχανικοί ίσω να μην είχαν μπορέσει να λύσουν τα προβλήματα σε αποθήκε αν δεν μπορούσαν να εργαστούν σε καταστάσει των πελατών τη εταιρεία του. Τώρα, διαδικασίε σε ό,τι αφορά το, η δοκιμή αγορά-εργασία. Η δοκιμή αγορά-εργασία θα καθυστερήσει δυστυχώ ε, ελπίζω θετική απόφαση για εφαρμογή αυτή της οδηγία. και κατά συνέπεια θα καθυστερήσει ή τέλο πάντων θα επιβραδύνει την δυνατότητα ε, παραδείγματο χάρη αυτών των ε, μηχανικών λογισμικού να πάνε στην Ισπανία και να λύσουν τα προβλήματα. Τέλο, αυτή η δωδεκάμινη περίοδος που προβλέπεται από την οδηγία είναι μακρά. Εγώ θα πρότεινα πιο μικρή χρονική περίοδο. Αν δούμε αυτά τα νεαρά στελέχη, παραδείγματο χάρη, που προσελήφθησαν να εργαστούν σε ξένε θεγατρικέ τη γερμανική μεταπητική βιομηχανή. Αυτά τα άτομα ήρθαν στην εταιρεία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά γρήγορα. Η περίοδο αυτή των 12 μηνών είναι πολύ μεγάλη και δεν θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην επιχείρηση αυτά τα στελέχη τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση. Άρα, ολοκληρώνοντα θέλω να πω ότι τα μέλη του Συμβουλίου μας ε, χαιρετίζουν τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων με Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο για την έγκριση τη οδηγία για τι ενδοϊπηρεσιακέ μεταθέσει, γιατί αυτό θα επιτρέψει δυναμικέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να, βελτι... να βελτιωθούν, αλλά θα βελτιώσει και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα που εξαρτάται τόσο πολύ από την ελεύθερη κυκλοφορία δεξιοτήτων και γνώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόξ. Τα όσα μας ήταν μια πολύ πρακτική εμπειρία. που μοιραστήκατε με τα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Αμέτ Νιφσαρκάρ. Νιφσαρκάρ, που είναι αντιπρόεδρος της ΝΑΣΚΟΜ. Ε, καλωσορίσατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή Λίμπε που με κάλεσε να δώσω την απόψή μου. Είμαι ο Αμέτε Νίβ Σαρκάρ, αντιπρόεδρος της ΝΑΣΚΟΜ. όσο δεν γνωρίζετε την ΝΑΣΚΟΜ, είναι μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις εργαζομένων στην, Ισλα... στην ε, Ινδία. Ε, είναι ε, ένας όμιλος τεχνολογικών εταιριών, ACB, Microsoft, έχουμε 1.300 εταιρείες, αλλά και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ινδία. HSBC, Philips, Siemens είναι και αυτές μέλη της, ε, του συνδέσμου μας. Έχουν εγκαταστήσει εκεί τα τμήματα τεχνολογικής ανάπτυξης, ε, στην Ινδία δηλαδή. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας κάνοντας μια σύντομη παρατήρηση γιατί υπάρχει ανάγκη για διεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια οδηγία όσον αφορά την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρειάζεται να διαχειριστούν ε, ε, πολλές δεξιότητες και προσόντα που υπάρχουν διαθέσιμα εκτός της Ευρώπης και είναι σημαντικό οι εταιρείε να είναι ευέλικτες και να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτές τις δεξιότητες, τα προσόντα σύντομα. Ε, πώς λειτουργεί στην πράξη. Μεγάλες, ας πούμε, μια μεγάλη εταιρεία Telecom έχει αναπτύξει μια νέα δυνατότητα για πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, σε πλατφόρμες όπως το iPad, ας πούμε. Στην πραγματική ζωή η λύση, ναι, αυτή η εξέλιξη αν ε, ε, έχει γίνει στην Ινδία και οι ψηλά ειδικευμένοι τεχνολο... Ε, τεχνικοί που δούλεψαν για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος πρέπει να μεταφερθούν, να ταξιδέψουν μάλλον στον πελάτη ούτω ώστε ο πελάτη να μπορεί να έχει την πρόσβαση στο σύστημα. Από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σύστημα, ο μηχανικό μετακινείται, πάει αλλού στον κόσμο ή αλλού ή επιστρέφει στην έδρα του. Είναι τόσο απλό. Όχι. Η Ευρώπη είναι μια ενιαία αγορά και αυτό ισχύει ίσως για τη μετακίνηση των προϊόντων, αλλά στις υπηρεσίες δεν είναι ακόμα ενιαία η αγορά για να σας ε, μιλήσουμε το ίδιο παράδειγμα. Αν αυτός ο μηχανικός ε, χρειαζόταν να έρθει σε τέσσερι διαφορετικές, ε, σε τέσσερις διαφορετικά μέρη σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα έπρεπε να πάρει ICT, άδεια εργασία, α πούμε, για τη Γερμανία, όταν θα έχει τελειώσει εκεί, να ξαναγυρίσει στη χώρα του, να πάρει μια νέα άδεια εργασία για τη Γαλλία, μόλι θα έχει τελειώσει εκεί τη δουλειά του, να ξαναγυρίσει στην Ινδία, να πάρει άλλη άδεια για τι κάτω χώρε και ούτω καθεξή, για να κάνει την ίδια εφαρμογή. Αυτό κοστίζει και καθυστερεί την εφαρμογή του προγράμματος. Και ποιος θα πληρώνει αυτό τελικά οι ευρωπαϊκές εταιρείες, ο ευρωπαίος καταναλωτής και οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες ε, διανύουν κρίση. Οι διάφορε χώρε έχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγηση, διαφορετικό χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση και τελικά αυτά προσθέτουν στην αβεβαιότητα του να εργάζεται κανεί στην Ευρώπη. Χρειάζεται εναρμονισμένη, απλοποιημένη, διαφανή διαδικασία, συνεπή διαδικασία για τι ε, μεταθέσεις αυτή τη αποσπάση, όπου θα επιτρέπει την ε, κινητικότητα μέσα στην Ευρώπη, επίση επαρκή ελέγχου, ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσει. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις γιατί έγιναν πολλές ερωτήσεις νωρίτερα για τις ε, διεπιχειρησιακές με αποσπάσεις. Τι δεν κάνουν αυτές οι αποσπάσεις. Ένα. Δεν είναι μόνιμη μετανάστευση. Έγινε μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έφτιαξε τη νέα, της πολιτική του πολιτική περιμετανάστευση, αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν για λιγότερο από 18 μήνε. Είναι άνθρωποι ειδικευμένοι, κάνουν μια δουλειά και μετά μετακινούνται στην επόμενη θέση του. Δεύτερον, αυτέ οι μετακινήσει δεν οφείλονται στην ανεργία. Ακούσαμε 16.000 μεταθέσεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και πάνω από ένα εκατομμύριο εργατικό δυναμικό είναι 0,2% του, του του, μάλλον του, του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Δεν θα επηρεάσει αυτό την ανεργία προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αντίθετα, θα βελτιώσει την καινοτομία και θα οδηγήσει έτσι στην ε, ευημερία και πιθανότατα μεγαλύτερη απασχόληση. Έπειτα, οι αποσπάσεις αυτές δεν είναι οι φθηνέ θέσει εργασία. Συχνά οι εταιρείε ψάχνουν να βρουν τοπικά το απαραίτητο προσωπικό. Και έτσι συνήθω λειτουργούν οι εταιρείε αυτέ. Πολλέ φορέ όμω οι ειδικοί, ιδιαίτερα οι πολύ ψηλά ειδικευμένοι, δεν υπάρχουν στην τοπική αγορά και γι' αυτό και του φέρνουν λόγω των γνώσεών τους. Σε περισσότερες περιπτώσεις το κόστος του να φέρει κάνει έναν ειδικό είναι ψηλότερο γιατί έχει το να πληρώσει το ταξίδι, τη, ε, τη στέγαση, τη, τα επιδόματα με την κατάσταση και ούτε καθεξής. Δεν είναι λοιπόν μόνιμη μετανάστευση, δεν οφείλεται στην ενεργεία και δεν είναι φθηνή εργασία οι αποσπασμένοι αυτοί άνθρωποι. Νομίζω πως το πεντάλεπτό μου τελείωσε τώρα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Now, we have heard... Ευχαριστούμε κύριε Νίβ Σαρκάρ. Ακούσαμε δύο εμπειρίες που σχετίζονται με το θέμα των διεπιχειρησιακών μεταθέσεων. Υπάρχει χώρος για συζήτηση για όσους θέλουν να κάνουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Κύριε Μούλντερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία πολύ σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Κόξ. Αυτή η περίοδος των 12 ε, μηνών ίσως θα πρέπει να θεωρηθεί και να ε, περιοριστεί. Επίσης, μήπως και η περίοδος των τριών ετών και αυτή να πρέπει να ε, συντμηθεί και αυτή ή είναι εντάξει αυτή η περίοδος αυτή. Κοιτάξτε, τα τρία χρόνια είναι η μέγιστη διάρκεια όπου ένας εργαζόμενος ICT μπορεί να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τρεις μήνες το ελάχιστο μέχρι σε τρία χρόνια το μέγιστο. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα, οι δύο παράμετροι που ορίζουν το πλαίσιο είναι ικανοποιητικοί. Συμφωνώ και εγώ ε, γιατί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους ICT δεν μένουν πάνω από 18 μήνες ή λιγότερο από 18 μήνες. For which Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τελικά μείναμε μέσα στο χρόνο μας, ε, στο χρόνο που είχε προβλεφτεί και αυτό μας ικανοποιεί. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι επιθυμούν ε, να φύγουν σήμερα το βράδυ για τις πατρίδες τους εγώ λοιπόν άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ε, παρεμβάσεις των ε, συναντέλφων που τοποθετήθηκαν σε αυτό που θα είναι η φάση επεξεργασίας του θέματος στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Άκουσα λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους εισηγητές ε, όλοι ανέφεραν ε, τεκμηριωμένες απόψεις ε, και την άποψή τους βέβαια για το θέμα που συζητάμε. Το θέμα αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και υπάρχουν ε, σημεία επαφής ε, με την ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Εκεί υπάρχει διαφορετική προσέγγιση από τη δική μου. Υπάρχει όμως, σας είπα, ένα σημείο επαφής και υπάρχει αρκετό περιθώριο έτσι ώστε ο καθένας ε, με τη δική την παρέμβαση να προσφέρει σε αυτό που νομίζει. Η σύνθεση θα είναι σύντομα απλή και σύντομη. Το έγγραφο αυτό επιθυμεί να προσφέρει υπεραξία το είπαν οι περισσότεροι. Υπεραξία στον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από εργαζόμενους που έχουν ιδιαίτερα προσόντα. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε άλλες μονάδες της ίδιας επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, από τη στιγμή που θα ε, γίνει αυτή η πρόταση οδηγία θα υπάρχουν ομοιογενείς, ενιαίες, ταχύες διαδικασίες Προηγουμένω, ο κύριο Κόξ είπε ότι υπάρχουν πολλέ δυσκολίε σε ορισμένε επιχειρήσει, γιατί οι επιχειρήσει δεν μπορούν χωρίς δυσκολία να επωφεληθούν νέου προσοντούχους ε, που θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμοι για μια εταιρεία. Ακούσαμε βέβαια και ε, αντίθετε απόψεις, απόψεις των ευρωβουλευτών, ακούσαμε τι ε, απόψει των εργαζομένων στον τομέα ε, ακούσαμε την άποψη της ε, κατηγορίας των εργαζομένων, ακούσαμε την άποψη των επιχειρήσεων, την άποψη εκείνου που θεωρεί ότι η πολιτική οικογένεια θα πρέπει και αυτή να ληφθεί επαρκώς υπόψη. Υπάρχουν ορισμένες ε, κατηγορίες εργαζομένων που υφίστανται ήδη, αλλά δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητος ορισμός. Οι ορισμοί θα πρέπει να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάποιος πρότεινε να υπάρχει και ως σημείο αναφοράς η συμφωνία GATS σε νομοθετικό επίπεδο. τι ε, ακριβώς ε, σημαίνει, ε, πώς ορίζεται ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ θα πρέπει να έχει την εξουσία, να έχει στη διάθεσή του ανθρώπινο δυναμικό, που να είναι μετρήσιμο, το οποίο, στο οποίο να μπορεί να ασκήσει το κύρος του. Δεν αρκεί δηλαδή να αναφερόμεθα μόνο στην ευελιξία, πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Κάποιος αναφέρθηκε στο άρθρο 14 και είπε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση ε, είναι καθοριστική βέβαια και ο πραγματικός στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τα νέα ταλέντα, την ε, ελευθερία εγκατάσταση και βέβαια και την επανένωση των οικογενειών. Γιατί αλλιώ δεν θα είναι ε, ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο, η μονάδα τη οικογένεια που μόλι συστήθηκε ε, αναγκαστεί να διαιρεθεί και πάλι. Εκπρόσωποι των εργαζομένων γυναικών μα είπε προηγουμένω ότι δεν πρέπει οι γυναίκες να παραμένουν στο σπίτι ενώ οι άνδρες εργάζονται. Άρα δηλαδή το θέμα της επανένωσης των οικογενειών πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι μεταναστευτικές ροές ε, είναι αχαλήνοτες ε, έγινε λόγος και για επανορισμό ε, της, ε, του του χώρου Σέγκεν. Εμείς θεωρούμε ότι τα κρατημέλη πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα και αυτό το συζητήσαμε και με το Συμβούλιο. ναι, νομίζω, ναι. Έγινε επίσης λόγος και για το χρονικό διάστημα για τους ε, υποδοκιμή εργαζόμενους. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη φάση και το είπαν αυτό αρκετοί εισηγητές, χρειάζεται μία επανένταξη ε, φρέσκων δυνάμεων, δυνάμεις οι οποίες βέβαια παράλληλα θα ενισχύονται από ένα ε, σωστό υπόβαθρο, από ε, πολιτιστικό κληροδότημα και από ουσιαστική γνώση. Μιλάμε δηλαδή για μεταφορά γνώσεων. Και έτσι ξεκίνησα και την δική μου την παρέμβαση. Είπα ότι πρέπει να καταστήσουμε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο ανταγωνιστικό, ένα σύστημα το οποίο θα ελκύει προσοντούχους ε, από άλλες ε, υπήρους, προσοντούχοι που θα έρθουν εδώ και θα εγκατσαθούν. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, οι μέθοδοι πρέπει να είναι απλουστευμένες και ε, ενιαίες. Όσοι προηγήθηκαν μου αναφέρθηκαν σε ένα πλαίσιο, σε ένα πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όπου θα πρέπει να εξαιρείται ο κατασκευαστικός τομέας. Εκείνο το οποίο πρέπει να δείτε σημασία είναι κυρίως τα δικαιώματα. Τα κοινωνικά θέματα είναι τόσο σημαντικά που αυτή η νομοθετική διαδικασία θα παρακολουθηθεί και από την ε, Επιτροπή Επασχόλησης. Είναι το πρώην άρθρο 50 για να δείξουμε ότι οι δύο επιτροπές ε, ενδιαφέρονται και οι δύο και είναι άμεσα υπεύθυνε για αυτή τη διαδικασία λήψης απόφασης. 16.500 ε, επιχειρήσεις μοιάζει να μην είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ε, παρόλα αυτά ε, θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε συζητήσαμε ταχύτατα και όσον αφορά στην ε, συμβολή, στη συνεισφορά που μπορεί να προσφερθεί στο μέλλον. Εμείς θεωρούμε ότι όσον αφορά αυτό το κείμενο και ε, εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάλεξε ε, για την παρέμβασή της. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παρουσιάσει σήμερα ε, αυτό το έγγραφο εργασία, το οποίο και προφανώ επιδέχεται βελτιώσει και βάσει όλων αυτών που ελέγχθησαν σήμερα εδώ. Στις 16 Ιουνίου αυτού του έτους ε, έχουμε καταληκτική ημερομηνία ε, για υποβολή τροπολογιών. Η συζήτηση θα γίνει Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου. Η πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή Επασχόλησης θα γίνει κατά την πρώτη ε, εβδομάδα του Οκτωβρίου, συγκεκριμένα στις 6 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία προς ανατολισμού στις 17 Οκτωβρίου ή τον επόμενο μήνα στις 23 ε, Νοεμβρίου. Θεωρούμε λοιπόν ε, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Πολωνική Προεδρία και σήμερα μίλησα με τον αρμόδιο Πολωνό Υπουργό ο οποίος είπε ότι επιθυμεί να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια με ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Η Πολωνική λοιπόν Προεδρία θα είναι ακριβώς εκείνη για να κλείσει ένα θέμα ε, που θεωρούμε όλοι ότι είναι απολύτως απαραίτητο και έτσι λοιπόν πέρα από τους ορισμούς ε, που περιλαμβάνει αυτό το θέμα, ένα άλλο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι εκείνο που έχει σχέση με τους εποχιακά εργαζόμενους. Πρόκειται για δύο θέματα που αλληλοσυμπληρώνονται. Ε, είναι θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις νόμιμες μεταναστευτικές ροές που και αυτές είναι άρρηκτα συνεδεμένες ε, με την αγορά εργασίας. Επειδή είμαστε πολύ κοντά στο Πάσχα θέλω να ευχηθώ σε όλους σας ε, ε, καλές γιορτές, καλό Πάσχα και ελπίζω ότι θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και με άλλους αδέλφους που για προφανείς λόγους δεν μπορούσαν να είναι παρόντες σήμερα εδώ. Πρόκειται για ένα θέμα ε, όπου κατά την άποψή μου είναι πραγματικά απαραίτητο να έχουμε σαφείς, ε, διαφανείς και αντικειμενικούς κανόνες. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο, κύριε Κόξ, ευχαριστώ όλους τους μετέχοντες, όλους όσοι ε, συμμετείχαν στο πάνελ και έκαναν ε, παρακολούθησαν αυτή την μακρά αλλά και χρήσιμη συζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι ε, η ανακεφαλαίωση που έγινε ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τις εργασίες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Μετά το Πάσχα και μετά από τις ε, ε, σύντομες αυτές ε, διακοπές ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν σας ευχόμαστε τα καλύτερα και ελπίζουμε ότι θα επανέλθετε με ανανεωμένη ενέργεια.